and we have a vote today. So, good morning. Good morning. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας στα αγγλικά, στα γαλλικά, ο πρόεδρος. Σας καλωσορίζω σε αυτή την τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών που έχει ως πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης την έγκρισή της με μια αλλαγή που θα ήθελα να σας επισημάνω. Η κυρία Γουξόμ που συμμετείχε σε μια αποστολή της αντιπροσωπείας στη Σικελία και θα μας κάνει μια ενημέρωση για αυτή την αποστολή. Πρότεινε να προσθεθεί αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη για να μας κάνει την ενημέρωση αυτής της επίσκεψης της αντιπροσωπείας μας στη Σικελία. Η ενημέρωση αυτή θα γίνει στις 5 που σημαίνει ότι οι συντονιστέ θα συνεδριάσουν γύρω στι 5.30. Θα ξεκινήσουν τη συνεδρίασή του γύρω στι 5.30 με την προσθήκη αυτού του νέου σημείου στην ημερήσια διάταξη. κυρία Βίξτρομ, λοιπόν, θα μα κάνει αυτή την ενημέρωση στι 5 το απόγευμα και οι συντονιστέ θα συνεδριάσουν από τι 5.30 και μετά. Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Να εγκρίνουμε και τα πρακτικά τη προηγούμενη συνεδρίαση. Αν δεν υπάρξουν ε, παρατηρήσεις ε, θα θεωρηθούν συγκεκριμένα και προχωράμε στο σημείο 4. Παρουσίαση από τον κύριο Wolfgang Goetz, τον οποίο και καλωσορίζουμε θερμά, τον ε, Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης ε, Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Θα μας ενημερώσει για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και της τοξικομανίας στην Ευρώπη με βάση τις μελέτη, τη μελέτη και την ετήσια έκθεση του 2010 από το Ευρωπαϊκό Αυτοκέντρο Παρακολούθησης. Καλωσορίζουμε τον κύριο Γκέτς, του δίνουμε το λόγο και κατόπιν θα γίνει συζήτηση. Κύριε Γκέτς, έχετε το λόγο. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με τα μεγάλη χαρά θα σας παρουσιάσω εδώ τα αποτελέσματα της μελέτης 2011 για τα προβλήματα της οξυκομανίας στην Ευρώπη αλλά τελικά θα ήθελα να σας πω ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις τις οποίες έχουμε λάβει μετά από την παρουσίαση στη Λισαβόνα στις 15 του Σεπτεμβρίου και ε, θα δείτε ότι αυτό το οποίο λάβαμε δεν είναι μόνο η έκθεση λάβατε δεν είναι μόνο η έκθεση είναι και πάρα πολλά επιμέρους θέματα άλλα στοιχεία και εθνικά προφίλ, δηλαδή η έκθεση δεν είναι ε, για μας μόνο μία έκθεση, είναι μία είσοδος επί της ουσίας σε ένα θέμα και είναι μία σειρά ενημερώσεων οι οποίες έχουν τοποθετηθεί στο διαδίκτυο και θα ενημερώνται συνεχώς. Και πρόκειται για μία έκθεση σχετικά με τις αντιθέσεις από τη μία πλευρά έχουμε ε, επίπεδα σταθερά ενώ υπάρχουν άλλοι τομείς όπως η χρήση κανάβεως από τους νέους που δείχνουν θετικές ε, αλλαγές. Αλλά η ε, εξέλιξη εις τα, τα συνθετικά ναρκωτικά και ο συνδυασμός ναρκωτικών με ινόπνευμα είναι ένα πολύ ουσιαστικό πρόβλημα και θεωρούμε ότι η Ευρώπη ε, έχει 1,3 εκατομμύρια τακτικών χρηστών και ενώ τα επίπεδα ήταν σταθερά μέχρι τώρα έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν όλο και περισσότεροι χρήστες που χρησιμοποιούν τις ενέσεις και υπάρχουν και υποκατάστατα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται ενεργά σε ορισμένες περιοχές. Ε, γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί διότι υπάρχουν πάρα πολλοί ε, οι οποίοι χρησιμοποιούν ε, θεραπείες υποκαταστάσεως αλλά ε, ε, και άλλες εξελίξεις ιδίως στις ανατολικές αγορές και βλέπουμε ότι στο τέλος του 2010 και αρχές του 2011 υπήρξε ε, μία εξέλιξη στον τομέα της χρήσεως ο ηρωίνης που οφείλεται ίσως στην καλλιέργεια του σχετικής ε, Παπαρούνας εις ε, την ε, στο Αφγανιστάν και ε, οδήγησε σε ορισμένες εξάρσεις ε, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με πάταξη ε, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών διότι με τα υποκατάστατα υπάρχει πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος θανάτου και είδαμε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, περίπου 7.500 περιπτώσεις οι οποίες μπόρεσαν να αποφευχθούν ε, και πέραν ε, των θανάτων υπάρχουν ε, τα δοτικές ασθένειες οι οποίες μπορούν να μεταδοθούν όπως άλλωστε και πολλές περιπτώσεις αυτοκτονιών και άλλες. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει πάταξη της χρήσης ναρκωτικών Ευρώπη και εδώ η έκθεσή μας καταλήγει στα εξή αποτελέσματα. Καταρχήν η πρόληψη του AIDS δεν ε, επιτυγχάνεται πάντοτε όσο θα θέλαμε και δεύτερον ξέρουμε ότι αυτή η ε, επιδημία πλήττει ιδιαίτερο σε ορισμένες χώρες και ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, οι υπηρεσίες πλέον δεν επαρκούν και λόγω της οικονομικής καταστάσεως διαπιστώνουμε και εδώ προβλήματα και βλέπουμε ότι στις ευάλωτες ε, κοινωνικές ομάδες υπάρχουν εξάρσεις. Η Ελλάδα παραδείγματος χάρη δήλωσε το ε, τελευταίο χρόνο παρόλα τα μέτρα ε, ότι αυξήθηκαν τα περιστατικά και τώρα τα ίδια στοιχεία με την Ελλάδα παρουσιάζουν και άλλες χώρες όπως παραδείγματος χάρη η Ρουμανία. Ας μιλήσουμε τώρα για το πιο σύνηθες ναρκωτικό που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη, την κάναβη, με πέραν του πολλών εκατομμυρίων χρήστες και βλέπουμε ότι όταν ενώ η χρήση είναι σταθερή ή μειώνεται σε ορισμένες χώρες πρέπει να μας ανησυχήσει η χρήση σε ορισμένες χώρες όπου είναι καθημερινή ε, και εκεί υπάρχουν περισσότερα προβλήματα από όσο όλοι οι άλλοι χρήστες συγκεντρωμένοι. Στην Ελλάδα παραδείγματος χάρη υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ζητούν βοήθεια και σε άλλες χώρες όμως. Και εδώ βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρξει μία επιλογή μεθόδων για να επηρεάσουμε τη χρήση και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία σαφής απόδειξη ότι μπορούμε να επηρεάσουμε το επίπεδο της χρήσεως κάναβης τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Υπάρχουν πιο περίπλοκοι παράγοντες που εμπλέκονται εδώ και θα χρειαστεί να σκεφτούμε πάρα πολύ καλά πώς θα χρησιμοποιήσουμε ε, τα φάρμακα που διαθέτουμε. Ε, πρόληψη ε, θα βασίζεται σε κοινωνικές προδιαγραφές και νομίζω ότι εκεί έχουμε κάνει μεγάλες προόδους. Παραγωγή της κανάβεως εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, είναι επίσης κάτι ανησυχητικό διότι το 2009 ε, έχουμε ε, κατάσχει 4,1 εκατομμύρια φυτά κανάβεως και μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κανάβεως κατάσχονται ετησίως διότι δηλαδή ε, ε, είναι προφανές ότι προσπαθεί κανείς να παράγει χωρίς να έχει διασυνοριακές συναλλαγές και ε, ακόμη και κοντά στις αστικές κοινότητες. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να αξιολογήσουμε ε, τη χρήση της κοκαίνης επίσης και είδαμε ότι 4,5 εκατομμύρια ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως χρησιμοποίησαν κοκαίνη πέρυσι και βλέπουμε ότι τα τελευταία στοιχεία παρουσιάζουν μία μείωση ενώ το θέμα της προμηθείας είναι λιγότερο σαφές και ε, η καθαρότης της ε, ποιότητας της κοκαίνης που διατίθεται έχει πέσει επίσης. Προσπαθούμε να ελέγξουμε την κατάσταση, ε, χρησιμοποιούμε μεθόδους πατάξεως αλλά βλέπουμε από τη μία πλευρά μία αύξηση χρήσεως παρόλο που προσπαθούμε ιδίω να πατάξουμε την, ε, το λαθρεμπόριο από τις χώρες της Αφρικής. Είδαμε ότι πέρυσι υπήρξε μία αύξηση κρίσεως των χαπακιών έκσταση τα οποία περιλαμβάνουν και άλλα ναρκωτικά όπως MCPP και αμφεταμίνες και ε, όπου υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και αυτό μπορεί να αναβιώσει το ενδιαφέρον στα χαπάκια αυτά έκσταση. Ε, είδαμε πέρυσι ότι είχαμε 41 επιπλέον νέες ουσίες οι οποίες επεσημάνθηκαν και φέτος ακόμη 39 πράγμα το οποίο δείχνει ότι στην αγορά εισάγονται συνεχώς νέα προϊόντα από την πλευρά της προσφοράς και μπορέσαμε να δούμε ότι στο διαδίκτυο που ολούνται πέραν των 600 προϊόντων και χρησιμοποιείται επίσης χρησιμοποιούνται και νέες ουσίες και γι' αυτό λόγω εξάρτησης ορισμένων ουσιών όπως το Μεθοντόλ το Συμβούλιο αποφάσισε να τοποθετηθούν και αυτά στον κατάλογο παρανόμων ουσιών αλλά το θέμα είναι πολύ περίπλοκο διότι υπάρχουν ε, πολλά ψυχότροπα, ε, ψυχότροπες ουσίες οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχούν ούτε στην Ευρώπη ούτε διεθνώς. Και προτού ολοκληρώσω κυρίες και κύριοι θα ήθελα να ε, εκφράσω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένες χώρες γιατί στο παρελθόν μόλις υπήρχαν προβλήματα μειωνόντουσαν ε, οι δαπάνες στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών πράγμα το οποίο επαναλαμβάνεται ε, τώρα και ε, σε περίοδο λιτότητος βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει να μας επισημάνει τα βασικά θέματα που προκύπτουν και για να μπορούμε να επενδύσουμε όπου η αποτελεσματικότητα θα είναι ε, εξακριβωμένη και πέρυσι είδαμε ότι παρουσιάστηκαν νέες ουσίες και του χρόνου θα είμαστε στην νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ε, ποια θα πρέπει να είναι η εικόνα της νέας στρατηγικής μας διότι μέχρι τούδε ε, μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε μία προσέγγιση η οποία ε, προσάρμοζε τις μεθόδους Ευρωπαϊκούς Ενώσεως της διεθνής αλλά τώρα όλες οι διεθνείς μέθοδοι συγκλίνουν και μπορούμε να μιλάμε για πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως το οποίο θα δώσει μια νέα όθηση για περαιτέρω σύγκληση και αυτό θα είναι ουσιαστικό για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στα ναρκωτικά και τη χρήση του στον 21ο αιώνα. Κυρίες και κύριοι, προσπάθησα να σας παρουσιάσω τα σημεία κλειδιά της στρατηγικής μας και πώς αντιδρούμε. Και πρέπει να πούμε ότι τα τα προγράμματα αυτά έχουν αλλάξει από ό,τι γνωρίζουμε και η αγορά των συνθετικών ουσιών στην Ευρώπη αλλάζει σημαντικά δηλαδή έσκασε η φούσκα της κοκαίνης και υπάρχει μία μείωση της καθαρότητας των χαπακιών ε, ε, έκσταση υπάρχει η αύξηση της χρήσεώς τους υπάρχουν νέες συνθετικές ουσίες που είναι διεγερτικά και όπως των το μεθατόν ε, μπορούν ε, να μετακυλήσουν από την νόμιμη στην παράνομη αγορά και θα δούμε ότι στο μέλλον θα υπάρξουν πολλές ουσίες που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο θέμα που μας απασχολεί αλλά τώρα μετά από την τελευταία δεκαετία προσπαθειών πρέπει να εξασφαλίσουμε την αντιμετώπιση των τωρινών και μελλοντικών προκλήσεων και θα ήθελα να τελειώσω αναφερόμενος εις ε, την ε, τελευταία έκθεση διότι παρουσίασε εμπιστευτικές πληροφορίες στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων και 15 Νοεμβρίου παρουσίασα το πρόγραμμα ή την Λισαβόνα όπου παρουσίασαν διάφορα κράτη-μέλη εθνικά προγράμματα που ξεκίνησαν. Έχουμε ε, τώρα το πρόγραμμα σε πάρα πολλές γλώσσες και ε, μπορεί κανείς να το κατεβάσει από το διαδίκτυο. Ε, είμαι λοιπόν ευτυχής ότι μέχρι στιγμής οι αντιδράσεις που είχα σχετικά με την ποιότητα του προγράμματός μας ήταν θετικές και όλοι είναι ευτυχείς ότι ε, υπήρξαν καλές αντιδράσεις διότι ουσιαστικά τα βασικά μας θέματα είναι τα νέα ναρκωτικά και η κοκαίνη και μετά από μία εβδομάδα είχαμε 1400 ε, νέα άρθρα και εκπομπές στην ε, τηλεόραση και εις ε, το ραδιόφωνο. Νομίζω ότι εφέτος θα φτάσουμε στις 3.000 διότι τα είχαμε ήδη προμίες εβδομάδος και ε, προσετέθηκαν η Κροατία, η Τουρκία και η Νορβηγία στο πρόγραμμα και ε, ξέρουμε ότι επίσης 150 αντιδράσεις υπάρχουν εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως στη Γερμανία και στην Ισπανία υπάρχει ενεργό ενδιαφέρον ε, μεγάλη κάλυψη σε επιπλέον στην Ρωσία, την Ελβετία, τις Ηνωμένε Πολιτείε και στην Κίνα, στην ε, Λατινική Αμερική, στη Βραζιλία και εδώ παρουσιάζω λίγα μόνο από τα στοιχεία των αντιδράσεων που είχαμε από όταν παρουσιάστηκαν αυτά τα προϊόντα και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας ε, ενδεχομένω σχετικά με τις αντιδράσεις αυτές. Σας λοιπόν- ευχαριστούμε κύριε Γκέτς. μπορούμε να συζητήσουμε την έκθεση. Ποιος θέλει το λόγο, ο κύριος είστε πρώτος. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον ε, Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για όλες τις πληροφορίες, τις πλούσιες πληροφορίες που μας έδωσε. Ως πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης ανησυχώ από τα στοιχεία που μας έδωσε ο κύριος Γκέτς. Και αν ήμουν ε, σε κυβερνών κόμμα ή συμμετείχα στην κυβέρνηση θα ήμουν ακόμη πιο ανήσυχο. Οι ε, κυβερνήσεις των χωρών μελών συνεργάζονται με το κέντρο σας και ποιες είναι οι αντιδράσεις ε, ε, απέναντι στην ετήσια έκθεσή σας. Επηρεάζει καθόλου η έκθεση αυτή τη διαμόρφωση των πολιτικών αυτών των κυβερνήσεων. Βλέπω ότι και η κυρία Τσίπελ ζήτησε το λόγο. Θεωρώ ότι η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που πρέπει να μας απασχολήσουν. Καταρχήν το θέμα του AIDS, διότι νομίζουμε, νομίζει η κοινή γνώμη ότι ε, δεν το ε, αντιμετωπίζουμε και η ιατρική ίσως υποδηλεί ότι ε, δεν χρειάζεται συνεχή επέμβαση, ενώ νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξαναεξετάσουμε από νέα σκοπιά και να δούμε ποιες είναι οι διαθέσιμες μέθοδοι. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι το θέμα του διαδικτύου σαν τρόπο αγοράς με απασχολεί και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει άμεση πώληση μέσω του διαδικτύου και αν υπάρχει διακίνηση εκεί και αν μπορέσει μπορέσει κανείς να προβεί σε έναν κατακαιρματισμό των διαφόρων μεθόδων. Ευχαριστώ. Η κυρία Φαγιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και το Διευθυντή του Κέντρου για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Έχω δύο ερωτήσεις ε, σύντομες. Καταρχήν για τις εθνικές στρατηγικές ε, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τοξικομανίας. Όπως ε, διαπιστώσαμε από την έκθεση, κάποιες χώρες έχουν ε, εθνικά σχέδια δράσης και εθνικές στρατηγικές, ενώ άλλες χώρες φαίνεται ότι υστερούν. Το 2011 έχουμε ακόμη χώρες μέλη που ε, δεν έχουν ετοιμάσει τέτοιες εθνικές στρατηγικές σχέδια δράσης. Και σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει δυστυχώς και η πατρίδα μου. Πώς σκοπεύετε να ασκήσετε πίεση ή υπάρχουν κάποιες προθεσμίες ε, που δεσμεύουν τους χώρες για να καταρτήσουν αυτές τις εκθέσεις ε, και να σας ενημερώνουν σε ό,τι αφορά την κάναβη. Πολύ ευαίσθητο αυτό το θέμα. Είναι από τα πιο δημοφιλή τέτοια παράνομα ναρκωτικά και δίστανται και απόψει ω προ το κατά πόσο θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση του ναρκωτικού αυτού. Πρόσφατα στη Σλοβενία διοργανώσαμε μία διάσκεψη και διαπιστώσαμε ότι οι νέοι είναι υπέρ της νομοποίησης ε, της κανάβεως. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη διάσταση και απόκληση και των πολιτικών, αλλά η δική σας γνώμη για την κάναβη ποια είναι, ποια πιστεύετε θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση της ε, κοινοτικής στρατηγικής για το τομέα αυτό. Άλλος κανείς? Ο κύριος Μπρόγκς. Πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο δεν έχουμε πρόβλημα, ένα ενιαίο πρόβλημα με τα ναρκωτικά, αλλά πολλά μικρά διακριτά πολλά ναρκωτικά επηρεάζουν τη συμπεριφορά ορισμένα από τα παρεστησιογόνα, μπορεί να προκαλέσουν διαεγκλήματα, εγκλήματα, αλλά απλά προκαλούν λίθαργο ή ε, μειωμένε ικανότητε κατά την οδήγηση. Αναφέρατε, υπάρχουν φυσικά συνέπειε για την υγεία, αλλά συνέπειε και για την εγκληματικότητα. Φυσικά, εάν μόνο για το έγκλημα θα μπορούσαμε να βρούμε πιο εύκολα λύσεις, αλλά υπάρχουν διάφοροι... Υπάρχουν δύο τρόποι προσέγγισης, η πλευρά ζήτησης και η πλευρά προμήθειας. Από την άψη της ζήτησης μπορούμε να έχουμε ένα γενικό μηχανισμό πυθού μέσω της ε, εκπαίδευσης, αλλά Επίσης ε, μπορείτε να γίνετε πιο πιστικοί όταν συγκεκριμένα άτομα συλλαμβάνονται από τις αρχές, ε, όταν καταλήγουν στη φυλακή. Από την από πλευρά της προμήθειας, ο κίνδυνος είναι ότι ε, αν αντιμετωπίσετε μόνο τους dealer μικρής κλίμακας ε, ε, που κάνουν χρήση σε σχέση με τους μεγάλες κλίμακας dealer που δεν κάνουν, χρήση, που κάνουν, που δεν κάνουν χρήση η συνέπεια θα είναι, οι συνέπειες θα είναι χειρότερες από ότι αν δεν είχατε παρέμβει καθόλου. Έτσι ε, το αποτέλεσμα θα είναι περισσότερες κλοπές ε, και περισσότερες ε, σε σπίτια και σε αυτοκίνητα. Ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε στον κύριο Γκέτς για να μας δώσει απαντήσεις για τα ερωτήματα που θέσατε. you uh, Ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που θέσατε. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε το βαθμό στον οποίο οι κυβερνήσεις ε, συνεργάζονται με το κέντρο παρακολούθησης για την πρόληψη των ναρκωτικών. Πρέπει να πω ότι το Διοικητικό Συμβουλίο μας, που είναι το σώμα που διοικεί την υπηρεσία, αποτελείται από αντιπροσώπους της κυβέρνησης, ε, κυβερνήσεων, μόνιμους αντιπροσώπους. Συνεργάζονται μαζί μας αποφασίζουν το πρόγραμμα εργασιών για παράδειγμα αλλά και για τα ζητήματα τα οποία θα εξετάσουμε πιο στενά Πρέπει επίση να τονίσουμε ότι η υπηρεσία μας δεν έχει πολιτική εντολή. Είμαστε ε, υπηρεσία πληροφοριών, παρέχουμε πληροφορίες, ενημέρωση και οι συνέπειες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους πολιτικούς, από όσους χαράσουν την πολιτική. Αυτό δεν εντάσσεται στι δικέ μα αρμοδιότητε. Έχουμε τακτικέ επισκέψει εκπροσώπων κυβερνήσεων σήμερα το απόγευμα. Έχουμε μια μεγάλη, ε, την επίσκεψη μια μεγάλη αντιπροσωπεία από το House of Lords, το Αγγλικό Κοινοβούλιο, και μερικές φορές ε, τέτοιοι άνθρωποι μα ζητούν πολύ συγκεκριμένε ε, πληροφορίε για συγκεκριμένες καταστάσεις στην Ευρώπη σε σχέση με τη διεθνή κατάσταση. Η αντιπροσωπεία αυτή του House of Lords θα έρθει για να σχηματίσει τη δική της γνώμη για το πώς θα μπορούσε να επηρεάσει τη στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα ε, αναπτυχθεί από το Συμβουλίο και την Κομισιόν μέσα στους επόμενους μήνες. Υπάρχει λοιπόν κάποια επιρροή αλλά δεν έχουμε άμεση επιρροή στο τι πράττουν οι κυβερνήσεις. Ε, κυρία Σίπλ, το HIV Äh, Αυτά μπορώ να τα πω γερμανικά εφόσον με ρώτησε γερμανίδιο. Σε μεγάλο, σε μεγάλο βαθμό έχει μειωθεί η πίεση και όντως πρέπει και εγώ να αναφερθώ στο θέμα των ε, μολύνσεων του AIDS ε, όσον αφορά τις άμεσες μολύνσεις διότι δεν μπορώ να αναφερθώ στη μετάθωση βλέπουμε ότι παραδοσιακά η Ελλάδα που ήταν μια χώρα με χαμηλό ποσοστό αλλά που τώρα είναι μια χώρα με πολλούς μετανάστες τα ποσοστά έχουν αυξηθεί και αυτό δεν σημαίνει ότι η μετανάστευση αυξίζει, αυξάνει τα ποσοστά του AIDS αλλά όταν έρχονται περισσότεροι σε ένα σημείο και οι υπηρεσίες που βρίσκονται εκεί είναι υπερφορτωμένες υπάρχουν και ανάγκες για επιπρόσθετο προσωπικό και αυτό αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Η Επιτροπή ΣΑΝΚΟ αυτή τη στιγμή εκδίδει μια προειδοποίηση σχετικά με το AIDS και ε, πρέπει να πούμε ότι έχουμε και το Ινστιτούτο για τις μεταδόσιμες ασθένειες στη Στοχόλμη και την Τετάρτη Πέμπτη νομίζω θα εκδοθεί ε, και την άλλη εβδομάδα θα δημοσιευθεί για την κατάσταση η οποία θα επισημαίνει και τον κίνδυνο για τη Βουλγαρία διότι και εκεί υπάρχουν όλο και περισσότεροι μετανάστες οι οποίοι ε, φτάνουν σε υπερφορτωμένες ορισμένες υπηρεσίες οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα τα περιστατικά όσον αφορά το θέμα των φαρμάκων τα οποία διακινούνται μέσω του διαδικτύου είπα ότι είχαμε διαπιστώσει στην, ε, στον τελευταίο απολογισμό τουλάχιστον 600 σημεία παραδόσεως ε, εις ε, την Ευρώπη ναρκωτικών σε 17 γλώσσες είχαμε κάνει απογραφές τον Ιανουάριο και και μετά τον Ιούλιο και αυτοί οι έμποροι στο διαδίκτυο προσπαθούν να βρίσκονται στο μετέχνιο μεταξύ νομιμότητος και παρανομίας. Βρίσκουν, ε, δεν θα βρείτε δηλαδή ηρωίνη και κοκαίνη αλλά χημικά παράγωγα ε, τα οποία είχαμε δει και την περασμένη εβδομάδα παραδείγματος χάρη συνθετικά καναβιοειδή και βλέπετε ότι οι έμποροι προσπαθούν να προστατευθούν διότι ε, ε, μέσως δίδουν και προειδοποιήσεις ότι κάτι μπορεί να είναι επικίνδυνο ή συνήθως σας παραπέμπουν ε, σε, ένα άλλο, σε μια άλλη ιστοσελίδα όπου είναι όμως τόσο περίπλοκο να φτάσετε που δεν θα διαβάσετε ποτέ τις προειδοποιήσεις και δεν είναι άτομα που βρίσκονται μόνιμα στο διαδίκτυο. Υπάρχει όπως είπα ένα μετέχμιο μεταξύ νομίμων φαρμάκων, παρανόμων ναρκωτικών, μία φεά περιοχή. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ουσίες οι οποίες είναι πολύ επικίνδυνες και πολλές φορές ε, δεν ε, λέγεται ε, όταν αγοράζετε αυτές τις ουσίες ποια είναι τα συστατικά τους όπως θα είναι η ε, το σούπερ μάρκετ. Επιστρέφω στα αγγλικά οι εθνικές ε, στρατηγικές ε, και έχουμε κάποια μείωση. Δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα η μείωσή τους, διότι αποτελεί γεγονός ότι πολλές από αυτές τις στρατηγικές και τα προγράμματα δράσης έχουν ε, δημιουργηθεί ταυτόχρονα και τώρα λήγουν σιγά σιγά σε όλες τις χώρες. Όλες οι χώρες προετοιμάζουν ήδη εθνικές στρατηγικές ε, και σχέδια δράση. Ε, φανταζόμαι λοιπόν ότι σε ένα χρόνο η κατάσταση θα είναι όπως πριν. Έχουμε σε όλα τα κράτη-μέλη μία επίσημη στρατηγική σχέδιο δράσης. Η μόνη χώρα που δεν έχει επίσημα ε, εγκεκριμένη στρατηγική είναι η Αυστρία. Αυτό όμως δεν είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί έχει περιφερειακές στρατηγικές και ε, τον εθνικό συντονισμό που τα διοργανώνει όλα αυτά. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να πω ότι η Αυστρία δεν έχει, γιατί σε κάθε περιφέρεια υπάρχει κάτι και υπάρχει ο εθνικό συντονισμό που τα συντονίζει όλα αυτά, αλλά δεν υπάρχει επισημοποιημένη ας πούμε, εθνική στρατηγική. Ε, τρόποι πίεση προ τι κυβερνήσει δεν έχουμε δυνατότητα να εξασκήσουμε πίεση σε κυβερνήσει. Ε, το όπλο μας είναι η ενημέρωση. Μπορούμε μόνο να παρουσιάσουμε την κατάσταση, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να εξασκήσουμε πίεση σε κανέναν. Αυτό είναι κάτι που ίσως να μπορεί να το καταφέρει καλύτερα η Κομισιόν, διότι η πλευρά της πολιτικής ορίζεται περισσότερο από την Κομισιόν, ε, ε, σχεδιάζεται από την Κομισιόν. Ε, ναι, άνθρωποι στη Σλοβενία και σε άλλες χώρες είναι υπέρ της νομιμοποίησης. Εάν είναι υπέρ της νομιμοποίησης, ε, προς το παρόν είναι παράνομη η κάναβης ε, σε όλα τα κράτη-μέλη. Αν θέλετε τη γνώμη μου, να σας πω την αλήθεια, δεν είναι δική μου δουλειά να σας δώσω τη γνώμη μου. Αν ε, πιούμε μια μπύρα μαζί μπορώ να σας δώσω τη γνώμη μου. μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρον να διαβάσετε την έκθεση της ε, Επιτροπής Κλωβή για τα Ναρκωτικά που είχε δημιουργηθεί από τον Μπάνκι και έχει περιλαμβάνει πολλούς πρώην αρχηγούς κρατών και αρχηγούς κυβερνήσεων και ο κ. Χαβία Σολάνα αποτελεί, ε, συμμετέχει σε αυτή την ομάδα. Πριν λίγες εβδομάδες δημοσίευσα μια έκθεση όπου δηλώνουν σαφώς ότι θα πρέπει να τα σκεφτούμε όλα, όλα τα ενδεχόμενα και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Όλες οι ιδεολογικές συζητήσεις έχουν εξαντληθεί, δεν κάνουμε πια ιδεολογικές ε, συζητήσεις. Αυτό που προτείνω πάντα στους πολιτικούς είναι να λαμβάνουν τα πάντα υπόψη και να εξετάζουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές ώστε να ε, διαπιστώσουν τι θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση. Συγγνώμη, ωστόσο δεν μπορώ να σας δώσω την προσωπική μου άποψη. Όσον αφορά τη δήλωσή σας, ε, ε, συμφωνώ μαζί σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκέτς. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή του τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας. Σας ευχαριστούμε και σας ε, ευχόμαστε ότι καλύτερα. Ευχαριστούμε για την επισκεψή σας. Θα σας ξαναδούμε και θα περάσουμε τώρα στο σημείο που φορά την τρομοποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών ή υπήκοοι των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου των τρίτων χωρών ή υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. η Εισηγητής ο κ. Ε, Διασδεμέρα. όπου εισάγονται οι νέες διατάξεις για διασφάλιση των θεωρήσεων για τις περιπτώσεις προσωρινής αναστολής ε, της απαλλαγής από για τρίτες χώρες. Θα ακούσουμε τον κύριο Διασδεμέρα και ίσως μετά τον αντιπροσώπο της Κομισιόν και την Πολωνική Προεδρία που ενδεχομένως θα είναι παρούσα στην αίθουσα ανακοινώνω ότι μετά από το επόμενο σημείο θα έχουμε ψηφοφορία. Όχι αυτό το σημείο, το επόμενο σας υπενθυμίζω λοιπόν να έχετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες ώστε να μπορέσουν, διαθέσιμες ώστε να μπορέσουμε να προβούμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία και όσοι από εσάς δεν τις έχετε φροντίσει να τις βρείτε. Για 10 λεπτά, εάν μου επιτρέπετε, θα μπορούσατε να προεδρεύσετε αυτό το σημείο. Η αντιπρόεδρος ε, της Επιτροπής Σοφιν Βέλ, επειδή έχω κάποια άλλη δέσμευση στην οποία θα πρέπει να ε, είμαι παρόν και θα επιστρέψω. Σε ευχαριστώ και θα επιστρέψω σε 10 λεπτά. Um, yes, I'm a bit unprepared. Good morning. Με βρήκατε απροετοίμαστη. Καλημέρα σας. Ας συνεχίσουμε τότε με την παρουσίαση της έκθεσης του κυρίου Δίας Δεμέρα. Θα ακούσουμε τον ε, εισηγητή. Πολύ καλημέρα σας και ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα αρχίσω την παρουσίασή μου εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου προς τους συναδέλφους ευρωβουλευτές, κυρίως τους κοιόδης συγητές, τα μέλη της Επιτροπής μας, αλλά και τους εκπροσώπους του Συμβουλίου για τη μεγάλη προθυμία τους, ε, την καλή προδιάθεσή τους και το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν μέχρι τώρα ε, για τη συζήτηση της τροποποίησης του κανονισμού 539 του 2001. Είναι η πρώτη φορά που εξετάζουμε αυτή την πρόταση κανονισμού και είναι η πρώτη φορά που θα σας εκφέρω και τη δική μου γνώμη ανεπιφύλακτα για το θέμα αυτό. Στις 20 Οκτωβρίου οι συγητές είχαμε μια συνεδρίαση, σύσκεψη με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής για να ενημερωθούμε διεξοδικά ε, για την κατάσταση και τις διάφορες πτυχές της πρότασης στην σύσκεψη αυτή, όπως θα, θυμάται και, θα θυμάται και η κυρία Φαγιόν. Μια στιγμή ε, διακόπτη πρόεδρος. Φαίνεται υπάρχει ένα πρόβλημα κάπου στα κανάλια της Δερμηνής. Συνεχίστε, συνεχίστε κύριε Σιγητά. Όπως έλεγα λοιπόν, στις 20 Οκτωβρίου ζήτησα από τους συναδέλφους να ξεκινήσουν ε, την κατάρτιση των τροπολογιών προκειμένου να διευκολύνουμε τη μελέτη του κειμένου και να έχουμε στενή συνεργασία και με την Πολωνική Προεδρία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας προτείνω λοιπόν για την υποβολή των τροπολογιών ε, τη Δευτέρα Δεκεμβρίου, μια πολύ ε, βραχία προθεσμία, αλλά έχω και δύο άλλες εναλλακτικές λύσεις, την 5η την 6η, 5η-6 Δεκεμβρίου γιατί πάνε περίπου 40 μέρε που ασχολούμαστε με τι τροπολογίε. Σα προτείνω λοιπόν τρει ημερομηνίε, 2, 5 και 6 Δεκεμβρίου. Ελπίζω να έχουμε έτοιμο τον κατάλογο πριν τι Χριστουγεννιάτικε διακοπέ αν τηρήσουν αυτές τι προθεσμίες. Ό,τι αφορά την ουσία της πρότασης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέραν κάποιων τεχνικών ζητημάτων, ε, η πρόταση αυτή έχει μια εξόχως πολιτική πρόταση και ένα εξόχως πολιτικό μέτρο, την λεγόμενη ρήτρα διασφάλισης, και τροποποιεί τον μηχανισμό της αμοιβαιότητας. Όπως είπα, η έκθεσή μου περιλαμβάνει 12 τροπολογίες. Θα αναφερθώ ξεχωριστά και απλά σε κάθε μία από αυτές. Η τροπολογία 1 προτείνει τροποποίηση του τίτλου του συγκεκριμένου θέματος της ρήτρα διασφάλισης. Εγώ προτείνω μηχανισμό ε, αναστολής προτιμώ αντί να λέμε ρήτρα διασφάλισης να μιλούμε για μηχανισμό αναστολής. Το ίδιο χαρακτήρα έχει και δεύτερη τροπολογία. Η τροπολογία 3 περιλαμβάνει μια πολιτική ε, δήλωση που ουσιαστικά ακολουθεί μια σύστηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, μια έντονη έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το οποίο ζητά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, εμπλέξει από τι αρχικέ φάσει τη διαδικασία με τη διαδικασία τη τροπολογία, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να προσκαλέσει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω προσκεκλημένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μην διαταράξουμε κανένα κανόνα. Η τροπολογία 4 ε, καθορίζει το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να επιλύει τι διαφορέ με βάση τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Η τροπολογία 5 είναι ένα θέμα συνοχή και συνέπεια. Αν θυμάστε, το Μάρτιο του 2011 ε, συντάξαμε δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού αμοιβαιότητα. Δηλαδή, αν με επιβραβεύσει, επιβραβεύω, αν επιβάλλει κυρώσει, το ίδιο και εγώ. Η τροπολογία 6 περιλαμβάνει τις το μηχανισμό αμοιβαιότητα που πρέπει να καλύπτει όλε τι περιπτώσει στι οποίε η αμοιβαιότητα δεν γίνεται σεβαστή. Τροπολογία 7 αφορά τι ε, ε, ε, δεσμεύσει που απορρέουν από διεθνεί συμφωνίε και τη δυνατότητα των κρατών μελών να απαλλάξουν από την υποχρέωση θεώρησης συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών. Καλό θα ήταν να διαγράψουμε την μία τρίτων, των υπηκών τρίτων χωρών. Λαμβάνοντα φυσικά υπόψη τη μελλοντική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι αποφεύγουμε νέες τροποποίησεις του κανονισμού γιατί μπορεί να ανακύψουν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη πρόταση τροποποίηση και φυσικά μιλάω για την Τουρκία όπως αντιλαμβάνεστε. Η τροπολογία 8 είναι πολύ συγκεκριμένη και θέλω να χρησιμοποιείται ο όρος ταξιδιωτικά έγγραφα και όχι άδειες διέλευσης, διπλωματικά ή υπηρεσιακά διαβατήρια και ούτω καθεξής. Ταξιδιωτικά έγγραφα να λέμε, για λόγους συνοχής. Ε, γιατί αυτό είναι, αυτή είναι η επίσημη ορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ταξιδιωτικά έγγραφα και είναι και μια ευρεία έννοια που καλύπτει όλους τους ε, τίτλους ταξιδιού και τα έγγραφα ταξιδιού. Τροπολογία 9. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα μέλη των πληρωμάτων της πολιτικής αεροπορίας εξαιρούνται μόνο κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν εξαιρούνται. Τροπολογία 10 και τροπολογία 11 που είναι και πιο ε, ουσιαστικές. Η τροπολογία 10 είναι και η πιο περίπλοκη από τις προηγούμενες γιατί προτείνει θέσπιση ενός γνήσιου μηχανισμού αμοιβαιότητας στις περιπτώσεις εκείνες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καταφέρει με διπλωματικά μέσα και τρόπους ε, μια τρίτη χώρα που τη χάνει εξαίρεση απαλλαγής να σταματήσει να απαιτεί αντίστοιχες ε, αξιώσεις από τους Ευρωπαίους πολίτες. Η περίπτωση του Καναδά δείχνει ότι παρά τις προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ισχύων μηχανισμός αμοιβαιότητας έχει σημαντικές αδυναμίες, χωλαίνει σε πολλά σημεία για ορισμένε χώρε μέλη. Γι' αυτό και θα πρέπει ο μηχανισμό αυτό τη αμοιβαιότητα να τροποποιηθεί. Επανεισαγωγή βέβαια τη υποχρέωση θεώρηση δεν γίνεται αυτόματα. Αλλά μπορεί να υιοθετηθεί προσωρινά αυτή η υποχρέωση μετά από μία ε, περίοδο διαπραγμάτευσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κράτους. Ε, μετά τι διαπραγματεύσει αυτέ, η Επιτροπή θα ενημερώνει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και σε περίπτωση που δεν ε, καταλήξει η συμφωνία Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την τρίτη χώρα, προτείνει ε, προσωρινή αναστολή που ε, θα εγκριθεί από κοινού από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Η εν λόγω απόφαση, και θα ήθελα να το διευκρινίσω, δεν επηρεάζει επουδενή το δικαίωμα πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ανά πάσα στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνεται να υποβάλει πρόταση τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού 539 κάθετος 2001. Γιατί εκεί κατα... περιλαμβάνονται οι πίνακες των χωρών που α, υπόκεινται ή όχι στην υποχρέωση θεώρησης. Και τώρα θα ήθελα να αναφερθώ διεξοδικά και πάλι στην τροπολογία 11. Αυτή αφορά την αναθεώρηση της ρήτρας διασφάλισης. Κατά τη γνώμη μου, ε, ε όρος ρήτρα διασφάλισης είναι αδόκιμος. Εγώ προτιμώ τον όρο ρήτρα αναστολής. Λοιπόν, ο μηχανισμός ε, της αναστολής που προτείνει σε κατάπικους περιπτώσεις, σε περίπτωση ε, κατάστασης που και αύξησης ε, των, των ροών. Τώρα, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι άσχετα με τους αριθμούς ή τα ποσοστά που θα συμπεριληφθούν τελικά στην πρόταση τροποποίησης του κανονισμού, τα ποσοστά αυτά και οι, αριθμοί απλώς ε, περιχαρακώνουν την διαδικασία αξιολόγησης, είναι δεικτικές. Θα εξαρτηθούν οι ειδικέ καταστάσεις ε, του ε, κράτους μέλους που πλήττεται και θα ληφθούν υπόψη οι εκθέσεις των αρμόδιων υπηρεσιών ή οργανισμών και εκεί θα αποφασιστεί αν θα δοθεί η αναστολή. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Ανάλογα με τις εκθέσεις θα ληφθεί η απόφαση για την αναστολή. Το γεγονός δηλαδή απλώς ότι φτάνουμε στα ποσοστά ή τους αριθμούς δεν αρκεί για να τεκμηριωθεί η αναστολή. Θα πρέπει επίση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερώνεται για οποιοδήποτε αίτηση αναστολής που έχει καταθέσει μια χώρα μέλος. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει, και το επισημένο θα συμμετάσχει έστω και ως προσκεκλημένο στη διαδικασία της επιτροπολογίας. Αυτό είναι κάτι που με βρίσκει σύμφωνο, αλλά είναι και το αποτέλεσμα των άτυπων συζητήσεων που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και χωρί να θέλουμε να παραβιάσουμε που δεν είναι τη διαδικασία τη επιτροπολογία. Απλώ θα προσκαλείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί έτσι υλοποιούνται και οι αρμοδιότητε και εξουσίε που προβλέπει η συνθήκη τη αναπόφαση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση τη διαδικασία τη. Ε, ε, με βάση τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Στην τροπολογία 11 προβλέπει τη δυνατότητα να χορηγηθεί εξαίρεση στα μέλη των σωστικών συνεργείων που σπέβδουν σε ένα κράτος μέλος σε περίπτωση θεομηνίας ε, ή ατυχήματος. Γιατί η πρόταση διαγραφής αυτής της κατηγορίας δεν έχει νόημα. Δεν θα απαιτήσουμε θεώρηση από το πλήρωμα ενός αεροσκάφους ε, που ε, σπέβδει να σώσει ε, Ανθρώπου που εξαιτία μια θεομηνίας βρίσκονται σε δινή κατάσταση. Έχουμε και την γνωμοδότηση τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που θα λάβω υπόψη. Ο συνάδελφος Κόβατσεφ προτείνει να ληφθεί υπόψη η έκθεση τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση πριν την ενεργοποίηση τη ρήτρα αυτή αναστολή, η ρήτρα διασφάλιση, όπω την αποκαλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί η ρήτρα αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει τι εξωτερικέ σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα μπορούσαμε να το διευκρινίσουμε ως εξής. Η... Λαμβάνονται υπόψη έκθεση της Frontex, της Europol, του, Ευρω... του Ευρωπαϊκού Γραφείου για το Άσυλο και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Αυτά κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σίγητα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Ντεκάιστερ για να σχολιάσει. Euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του όπου αναφέρονται τροπολογίες αυτού του κανονισμού 539 και οι διατάξεις για την πολιτική για τις θεωρήσεις στο γενικό πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την πρόταση της Κομισιόν έχουν γίνει πολλές τροπολογίες που θα χαρακτηρίζαμε μάλλον τεχνικές αλλά υπάρχουν και ορισμένες που πράγματι θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης. Σε αυτή μου την ομιλία θα ήθελα να επικεντρωθώ πρώτα απ' όλα στα σημαντικότερα σημεία στις ε, προτάσεις τροπολογιών του εισηγητή σε σχέση με τις ρήτρε διασφάλισης, σε σχέση με το μηχανισμό αναστολής, το απαλλαγής αποθεωρήσεις και για τη ρήτρα του μηχανισμού αμοιβαιότητα. Γενικά η Κομισιόν ε, επικροτεί αυτό το σχέδιο έκθεση και τι τροπολογίες θεωρούμε ότι οι περισσότερες τροπολογίε ευθυγραμμίζονται με τι αρχέ που υποστηρίζουν την πρόταση της ε, Κομισιόν αλλά τη βελτιώνουν σε κάποια σημεία με μία ίσως εξαίρεση της τροπολογίας σε σχέση με το μηχανισμό αμοιβαιότητας αλλά θα επανέλθω σε αυτό. Όσον αφορά ορισμένες μάλλον τεχνικές τροπολογίες όπως για παράδειγμα η απαλλαγή αποθεωρήσεις για τα μέλη μη στρατιωτικών πληρωμάτων αεροσκαφών μπορούμε να αποδεχθούμε αυτή την τροπολογία η οποία διευκρινίζει ότι αυτή η απαλλαγή από θεωρήσεις εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που αυτά τα μέλη πληρώματος ε, εργάζονται και όχι όταν πάνε διακοπές. Αυτή είναι μια διευκρίνηση φυσικά αλλά ε, συμφωνεί με την αρχική ιδέα της Κομισιόν. Όσον αφορά τη ρήτρα διασφάλισης ή το μηχανισμό αναστολής των θεωρήσεων, για να ανταποκριθούμε σε περίπτωση εκτακτής ανάγκης, σε περιπτώσεις κρίσης, η Κομισιόν πρότεινε να ε, προσφύγουμε σε μια διαδικασία επιτροπολογίας ώστε να εγκριθεί ενδεχομένως μια απόφαση με την οποία αναστέλλεται η απαλλαγή αποθεωρήσεις ε, που έχει χορηγηθεί σε μια τρίτη χώρα. Για εμάς αυτή είναι η μόνη διαδικασία που μας επιτρέπει γρήγορη αντίδραση. Προφανώς, εάν θέλουμε να προχωρήσουμε στο πλαίσιο της επιτροπολογίας, τα κριτήρια που επιτρέπουν την ενεργοποίηση της διαδικασίας θα πρέπει να έχουν καθοριστεί με σαφήνεια. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν ασαφή κριτήρια τα οποία επιτρέπουν μεγάλο περιθώριο εκτίμηση στα κράτη-μέλη για την ενεργοποίηση του μηχανισμού και για την Επιτροπή, για την Κομισιόν όταν πρέπει να λάβει θέση για το ζήτημα του κατά πόσο πρέπει να ανασταλεί ή όχι η απαλλαγή από θεωρήσεις. Για αυτό το λόγο στην πρότασή της η Κομισιόν έχει ορίσει κριτήρια, θα έλεγα μαθηματικά, τα οποία ε, δεν ε, αφήνουν ε, ιδιαίτερες ελευθερίες αυθαίρετες. Η Προεδρία θα μας εξηγήσει σε λίγο ότι στο Συμβουλίο τα κρατημέλη είναι μάλλον υπέρ πιο ασαφών κριτηρίων που επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία ενώ ταυτόχρονα θέλουν να καθοριστούν κριτήρια στην Κομισιόν όταν προετοιμάζει την ενδεχόμενη αναστολή της απαλλαγής από Η Κομισιόν έχει σημειώσει τις ε, τροπολογίες του εισηγητή, ο οποίος ε, συνεχίζει να εργάζεται με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά είναι βέβαιο ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες ε, θα γίνουν αρκετές συζητήσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και εκεί η Κομισιόν θα έχει την ευκαιρία να επανεξετάσει ή να προσαρμόσει τη θέση της σε συνάρτηση με τις απόψεις που θα εκφράσουν τα άλλα δύο όργανα. Ο μηχανισμός αμοιβαιότητας τώρα, η Κομισιόν είχε προτείνει την τροποποίηση του υπάρχοντος μηχανισμού σε ένα μόνο σημείο, δηλαδή ευθυγράμμιση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η Κομισιόν, ωστόσο, είχε πει από την αρχή ότι ήταν διατεθειμένη να ακούσει τις ε, πιθανές, ε, όποιες τυχόν προτάσεις, βελτίωσης του μηχανισμού, προτάσεις, συστάσεις που θα μπορούσαν να καταστήσουν πιο αποτελεσματικό τον υπάρχοντα μηχανισμό. Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε τις ε, προτάσεις του εισηγητή. Φυσικά θα πρέπει ούτως ή άλλως να φροντίσουμε αυτές οι βελτιώσεις να λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο που ορίζουν οι συνθήκες. Επ' αυτού θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε τη συζήτηση. Επ' αυτού λοιπόν η πρόταση που κάνει ο εισηγητή για επιβολή στην Κομισιόν μια υποχρέωση μετά από 90 ημέρες, μετά από τη δημοσίευση ε, της ενεργοποίησης του μηχανισμού αμοιβαιότητας να υπάρξει πρόταση που αποσκοπεί στην απαλλαγή από τις θεωρήσεις μας φαίνεται πιο συμβατό με το δικαίωμα, αποκλειστικό δικαίωμα πρωτοβουλίας της Κομισιόν. Δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο ελευθερίας εκτίμησης στην Κομισιόν να υποβάλει ή όχι πρόταση. Εδώ λοιπόν διατηρούμε ένα ερωτηματικό εμείς ως Κομισιόν αυτό το τμήμα της τροπολογίας ε, που προτείνει ο εισηγητής. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι από την αρχή η οχι προταση εδω λοιπον διατηρουμε ενα ερωτηματικο εμεις κομισιον αυτο το τμημα της τροπολογιας που προτεινει ο εισηγητης σε αυτο το πλαισιο θα ηθελα επισης να υπενθυμισω οτι απο την αρχη η κομισιον είπε ότι αυτό είναι ένα πολιτικά πολύ σημαντικό και ευαίσθητο θέμα. Θα πρέπει να δούμε επίσης πώς μπορούμε να το συζητήσουμε με το Κοινοβούλιο σε περιπτώσεις ε, τέτοιων προβλημάτων. Εδώ επανέρχομαι στη ρήτρα διασφάλισης ε, αλλά και για τα δύο ισχύει αυτό. Η ρήτρα διασφάλισης ε, αποσκοπεί σε μια ενδεχόμενη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της επιτροπολογίας. Εκεί φυσικά τίθεται ένα μικρό πρόβλημα. Είμαστε έτοιμοι να εμπλέξουμε περισσότερο το Κοινοβούλιο, ωστόσο θα πρέπει να σεβαστούμε τους κανόνες της επιτροπολογίας όπως έχουν συμφωνήθει μεταξύ των οργάνων. Αυτά κυρία Πρόεδρε θεωρώ ότι ήταν τα σημαντικά μου σημεία των αρχικών αντιδράσεων στο σχέδιο τροπολογιών Φυσικά είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε περισσότερες εξηγήσεις για τα πιο τεχνικά σημεία. Καλώς. Ξαναδίνω την Προεδρία στον κύριο Αγγιλάρ. Yes. so much. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, κυρία Σόφι Εντβέλτ. Ε, με αναπληρώσατε όσο εκπλήρωνα την άλλη ενηλειμμένη μου υποχρέωση. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Προεδρία του Συμβουλίου ε, στον κύριο Φιλίπ Ζαζίνσκι. Καλημέρα σας και καλημέρα κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου ε, για τις θεωρήσεις δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο σημαντικό θέμα επιτάπητος και θα ήθελα να είμαι ειλικρινής απέναντι σας ε, απέναντι στα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Ακόμη και πριν ε, λάβουμε το κείμενο της έκθεσης, ε, σε κάθε συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας και της Θεωρήσης είχαμε ενημέρωση των αντιπροσωπιών ε, για να εξοικειωθούν με τις αρχικές παρατηρήσεις και την προκατακτική προσέγγιση των μελών της Επιτροπής σας. Και σας διαβεβαιώ ότι τα μέλη της ομάδας εργασίας για τις θεωρήσεις ε, άκουσαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις και θέλουν να βρουν ε, όσο δυνατόν μεγαλύτερη ισορροπία και σύγκληση μεταξύ των ε, απόψεων του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Και θα ήθελα να εκφράσω την μεγάλη μου ευγνωμοσύνη προς τον εισηγητή τον κύριο Δία Δεμέρα για την προθυμία και το πνεύμα συνεργασία που έδειξε απέναντι στο Συμβούλιο. Γιατί εμείς από το πρώιμο στάδιο τη Διαδικασία φροντίσαμε να έρθουμε σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ενημερωθούμε για τις απόψει του. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη ελπίδα για ανέβρεση λύσης. Γιατί διαβάζοντας την έκθεση του κυρίου Δίας Δεμέρα, διαπιστώνω ότι κάνω δύο σημεία μόνο χρήζω διευκρίνησης. Το πιο σημαντικό όμως είναι και χαίρομαι που το ανακοινώνω. Βέβαια, όχι, δεν χαίρομαι γιατί διαφορούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι όμως που τουλάχιστον τα ε, μέλη της Ομάδας Εργασίας ε, για τις Θεωρίες του Συμβουλίου αντιλαμβάνονται ότι όταν μιλάμε για ρήτρα διασφάλιση ή μηχανισμό αναστολή, όπω και να τον αποκαλέσουμε τελικά, το, ε, το εργαλείο αυτό θα πρέπει να είναι ε, σωστό και υγιέ. Γιατί όταν ενεργοποιείται το εργαλείο αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο που δεν θα είναι αυτόματο. ούτε θα επιτρέπει διακριτική μεταχείριση και αυτό θα πρέπει να αποσαφηνίζεται στον κανονισμό. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέλο στο Συμβούλιο που να διαφωνεί με αυτή την άποψη. Παρ' όλα αυτά, το μείζον πρόβλημα, και τώρα θα ήθελα να επικεντρωθώ στο μηχανισμό της αναστολής, γιατί θα ήθελα να επισημάνω ότι τα υπόλοιπα σημεία σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, δεν μας ε, χωρίζουν. Η μόνη εξαίρεση ίσως είναι η συζήτηση για την αμοιβαιότητα, γιατί δεν έχει γίνει ακόμη στο Συμβούλιο η συζήτηση για την αμοιβαιότητα. Είμαστε σε φάση ε, προκαταρκτική ακόμη για την αμοιβαιότητα. Για τον μηχανισμό αναστολής πάντω ήθελα να είμαι σαφής. Αν εφαρμόσουμε μία αμυγή μαθηματική προσέγγιση στην ε, άκρος πολιτική και πολύ σημαντική ε, λύση, τότε θα πρέπει να γυρίσουμε στα θρανία και στα μαθήματα μαθηματικής, μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο. Αυτό όμως δείχνει ότι δεν αναγνωρίζουμε και δεν αντιλαμβανόμαστε τα περίπλοκα πολιτικά ζητήματα. Το Συμβούλιο θέλει να κρατήσει τα ποσοστά ως επικουρικό όμως μέσο για την αξιολόγηση της κατάστασης. Αυτό που κάνει το Συμβούλιο και αυτό που προτείνει και η Πολωνική Προεδρία και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει είναι να δώσουμε εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αρμοδιότητα να αξιολογήσει τις λεπτομερείς πληροφορίες του κράτους μέρους που αντιμετωπίζει προβλήματα και να διαπιστώσει κατά πόσο οι ανακοινώσει που έγιναν και οι πληροφορίες που δόθηκαν από το κράτος μέλος είναι έγκυρες. Και από τη στιγμή που γίνει αυτή η κοινοποίηση, ε, θα ξέρουμε περισσότερες θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες ε, ε, για συγκεκριμένους το δυσάσυλο, αλλά η προσέγγιση μας δεν θα είναι αμυγός μαθηματική, θα είναι πιο πολιτική. Και σε αυτή τη φάση της διαδικασίας θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη πολλές πληροφορίες από την έκθεση Frontex, από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ακόμη και από την έκθεση της Europol. Αυτό δεν σημαίνει ε, ότι θα πρέπει να γίνεται σίγουρα μία στο οργανωμένο έγκλημα. Ήδη αυτό το κριτήριο υπάρχει και στο πρώτο σκέλος του μηχανισμού. Πάντως, το βασικό μήνυμα που θα ήθελα να απευθύνω στην Επιτροπή σας, στην Επιτροπή Πολιτικών ελευθεριών είναι αυτή τη στιγμή υπάρχει σαφής συμφωνία και αντίληψη ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα ίδια κριτήρια όταν αξιολογούμε την κατάσταση στη Γερμανία ή το Λουξεμβούργο. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια κριτήρια εφαρμόζοντας τη ρήτρα αυτή προς οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Γιατί υπάρχουν διαφορές και αυτό που προτείνουμε είναι να αναλάβει μεγαλύτερη πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει ε, διεξοδικά και ευρυθώς ε, περιπτωσιολογικά το κάθε δοσία και να μην εφαρμόζει μαθηματικά και ψυχρά την προσέγγιση αυτή. Αυτή είναι η στάση του Συμβουλίου. Κυρίε και κύριοι, και σα διαβεβαιώ ότι θέλουμε η διαδικασία να γίνει πιο ελαστική, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανελαστικότητα και θέλουμε να την καταστήσουμε και πιο αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τζαζίνσκι. Στρέφουμε τώρα προ τα μέλη τη Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών. Ε, θα λάβει πρώτα το λόγο η κυρία Φαγιόν που είναι και σκιώδη συγγήτρια για το θέμα αυτό. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και το Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς άλλωστε και τους άλλους σκιώδης εισηγητές ε, για τα σχόλια διότι θα ήθελα να σας πω ότι καταρχήν είμαι πολύ ευτυχής με τις προτάσεις και πιστεύω ότι οι τροπολογίες είναι πολύ καλές, ε, βελτιώνουν το κείμενο και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε καλές λύσεις στο τέλος. Όσον αφορά ε, τα, ε, την προθεσμία για τις τροπολογίες νομίζω ότι είναι 5 ή 6 Δεκεμβρίου διότι 2 Δεκεμβρίου είναι ήδη αυτή την εβδομάδα και την ε, περασμένη εβδομάδα είχαμε εκλογέ στη Σλοβενία οπότε ήδη είχα πρημοδοτήσει την επόμενη εβδομάδα και φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει προβλήματα. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες και θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένες από αυτές όσον αφορά την ρήτρα διαφυγής για τις θεωρήσεις πιστεύω ότι δεν είναι σωστός όρος ο υπάρχει καλύτερος όρος να μιλάμε όχι για ρήτρα αλλά για μηχανισμό ε, και ε, νομίζω ότι αυτή θα ήταν η σωστή, ε, ο σωστός χαρακτηρισμός. Επίσης όσον αφορά τον ρόλο του Κοινοβουλίου που έχουμε υπάρξει θετική στο παρελθόν στο ρόλο του Κοινοβουλίου και νομίζω ότι θα πρέπει να βαθμιστεί ο ρόλος αυτός ήδη στην αρχή της επιτροπολογίας. Ήμουν σκιώδης εισηγήτρια όταν προτείναμε και στηριχθήκαμε σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να υποβάλει την πρότασή του πριν από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, ελπίζω ότι αυτό δεν είναι ένα αρνητικό βήμα για την Επιτροπολογία και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αντιληφθεί ε, πώς έχει κατάσταση και θα έχει έναν επικοδομητικό ρόλο από την αρχή αρχή. Βεβαίως δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με την ανάγκη αμφίδρομης λειτουργίας και θα έλεγα να στηριχθεί ο μηχανισμός αυτός αλλά χρειάζονται βελτιώσεις για να καταλήξουμε σε μια κοινή οδό όπου θα συμπλέψουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Συμβούλιο και πιστεύω ότι το πιο βασικό είναι ίσως οι αριθμοί διότι παρόλα αυτά Χαιρετίζω την πρόταση του Συμβουλίου ότι δεν πρέπει αυτό να αποτελέσει το βασικό κριτήριο διότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έχει αναφερθεί σε την διαγραφή των ποσοστών αλλά εμείς θα έπρεπε ίσως ε, να αναφερόμαστε εις ε, ε, μία εξαιρετική ή υπερβολική αύξηση ετούντων άσυλο που θα επηρέαζε την μεταναστευτική εικόνα σε αυτή τη χώρα και αυτό το έχουμε διαπιστώσει όχι μόνο στην προηγούμενη χρονική περίοδο αλλά σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η πρόθεση ε, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να χρησιμοποιήσουν άλλους μηχανισμούς χωρίς όμως να αποφύγει κανείς το γεγονός ότι ο νέος κανονισμός αυτός δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αριθμητικά και θα πρέπει ε, οι αριθμοί να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι διαφαίνεται στην αρχή της προσπαθίας. Στηρίζω λοιπόν την πρόταση του εισηγητή και προσωπικά δεν πρόκειται να διατυπώσω άλλες τροπολογίες και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μία ε, ισοσκελισμένη αντιμετώπιση από τα διάφορα θεσμικά όργανα κατά τρόπον ώστε να ικανοποιηθούν και τα κράτη-μέλη. Η ισχυώδηση συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μερικά σχόλια. Εδώ μιλάμε για μια τεχνική έκθεση με τεράστιο πολιτικό ενδιαφέρον και τεράστιε πολιτικέ συνέπειε. Η αλήθεια είναι ότι ω εκπρόσωποι των πολιτών μας ε, σίγουρα θα πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα την ε, ευαισθησία του θέματος, ειδικότερα όσον αφορά τα ταξίδια εκτός του χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προβλημάτων που υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. τα τελευταία δέκα χρόνια είχα αλλάξει περίπου δέκα διαβατήρια για διάφορους, ε, λόγω διαφόρων απαιτήσεων ε, θεωρείς, για θεωρήσεις και γι' αυτό έχω κάποια ευαισθησία για αυτό το θέμα. Ε, σε μια ιδανική Ευρωπαϊκή Ένωση, αλληλεγγύη, θα πρέπει να αποτελεί κυριαρχή μεταξύ μας, αλλά δεν ζούμε σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε να φτάσουμε εκεί κάποια στιγμή, κάποια χρονική στιγμή, αλλά ε, την παρούσα στιγμή δεν υπάρχει αλληλεγγύη για παράδειγμα όταν μιλάμε για τρίτες χώρες που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη ακόμη και η λέξη κράτη-μέλη κάποιου πράγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ζήτημα έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά τις σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες Φυσικά η αλληλεγγύη συνεπαγέται επίση λογικά ότι αφού ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της θα έπρεπε να απαντήσει αλλά όπως είπα η αλληλεγγύη δεν αποτελεί ακόμα πραγματικότητα εάν ελπίζουμε ότι κάποτε θα το αποτελέσει πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο στον πραγματικό κόσμο στον οποίο ζούμε για να δούμε πόσα μπορούμε να επιτύχουμε υπό αυτές τις συνθήκες. Ανεξάρτητα ίσως από το γεγονός ότι πραγματικά πολύ πρόσφατα μία δήλωση ψηφίστηκε από την πλειοψηφία αυτού του κοινοβουλίου που, την οποία απαιτήθηκε αυτή η αρχή αλληλεγγύης να είναι παρούσα. Επειδή πρόκειται για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες, με χαρά λέω ότι είμαι ευχαριστημένη που ο εισηγητής ε, αυτού, αυτής της έκθεσης, ο φίλος μου, ο κύριος Αγκουστίνδιας Δεμέρα, έχει καταφέρει με έναν πολύ ισορροπημένο και λογικό τρόπο να αντιμετωπίσει την κατάσταση και κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο υπό τις ε, τρέχουσες θήκες. Ε, όπως έχουν λοιπόν τα πράγματα αυτή τη στιγμή θα περιοριστώ σε μόλις δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι ότι θα ήθελα να καταλάβω αυτή η αλλαγή από το 50% στο 60% για να μπορέσουμε να κρίνουμε κατά πόσο το 60% είναι το σωστό ποσοστό. Ποιος είναι ο λόγος ε, για τον οποίο περνάμε από το, 60, από το 50% στο 60%. Και η άλλη μου ερώτηση σχετίζεται με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπολογία. Θα ήθελα να καταλάβω πώς αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει πρακτικά, τι είδους διαδικασίες απαιτούνται, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντίθετα από τα Εθνικά Κοινοβούλια, έχει, εργάζεται διαφορετικά όπως για παράδειγμα κατά τις καλοκαιρινές διακοπές, τις πράσινες εβδομάδες, τις χειμερινές διακοπές δηλαδή θέλω να μιλήσω τεχνικά θέλω να ρωτήσω πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτι τέτοιο πρακτικά Όσον αφορά τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ξέρω, έως την προθεσμία υποβολή των τροπολογιών ίσως και εγώ να σκεφτώ κάποια τροπολογία η οποία θα μπορούσε να μας δώσει ας πούμε περισσότερη εξουσία περισσότερες δυνατότητες ευχαριστώ Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουσουτήλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ μαζί με τους συναδέλφους να συγχαρώ θερμά τον κύριο Δίας Δεμέρα για την έκθεσή του, για την παρουσίαση που μας έκανε σήμερα και την κατάθεση των τροπολογιών του. Και εγώ πιστεύω ότι αν θέλουμε το καθεστώς των θεωρήσεών μας να είναι αξιόπιστο, είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε και ένα μηχανι... έναν αποτελεσματικό μηχανισμό αναστολής που θα λειτουργεί όταν γίνεται κατάχρηση του συστήματος των θεωρήσεων και είναι σημαντικό αυτό το μήνυμα να το μεταφέρουμε στους πολίτες. Δηλαδή δεν θέλουμε απλώς να διευκολύνουμε την απαλλαγή των θεωρήσεων, φυσικά αυτό είναι καλό, αλλά είμαστε ικανοί ακόμη και να αναστείλουμε ε, το σύστημα αυτό, αν διαπιστώσουμε ότι λαμβάνει η χώρα κάποια κατάχρηση του συστήματος ε, απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Θα ήθελα να υποβάλω δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τον εισηγητή. Ε, η πρώτη ερώτηση είναι χρονική, χρονικού ορίζοντα. Τι χρονοδιάγραμμα έχετε υπόψη σε ό,τι αφορά την ε, δημιουργία μιας κατάστασης ε, που υπάρχει πιθανότητα κατάχρησης μέχρι τη λήψη της, αποτελεσματικής, της απόφασης για την, για την εφαρμογή του μηχανισμού αναστολής και ε, για το δεύτερο θέμα που έδειξε το Συμβούλιο. Ποια είναι η γνώμη του εισηγητού ε, για τη διαφοροποίηση. Γιατί όπως είπε το Συμβούλιο, άλλο η κατάχρηση να επηρεάζει το Λουξεμβούργο και άλλο οι μετανάστες πηγαίνουν προς τη Γερμανία. Γιατί εκεί θα είναι διαφορετικός ο αντίκτυπος, πιο δύσκολος. Η κατάσταση κατάχρηση μιας χώρας που αισθάνεται ότι έχει κατακλειστεί από το φαινόμενο αυτό θα λαμβάνετε υπόψη για τη χρήση του μηχανισμού αναστολής από την απαλλαγή Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κυρία Τσίπελ. Ευχαριστώ. Έχω μόνο μία πολύ σύντομη ερώτηση ε, για ένα πρόβλημα που αντιμετώπισα τις τελευταίες μέρες και δεν ξέρω αν αυτό έχει σημασία στις συζητήσεις διότι καταρχήν υπάρχει ο κατάλογος των χωρών που μπορούν να ταξιδεύσουν χωρίς θεώρηση και ε, μία, ένα δεύτερο κατάλογο ε, ασφαλών τρίτων χωρών όπως ονομάζονται και οι πολίτες αυτοί μπορούν να ταξιδεύσουν χωρίς θεώρηση σαν τουρίστες και στο τέλος ζητήσουν, ζητούν άσυλο αλλά εάν, ε, ε, εάν στο τέλος του, της παραμονής αυτής τους αρνηθούν αυτό το άσυλο δεν μπορούν να τους αποστείλουν στη χώρα προελεύσεώς τους διότι δεν θεωρείται ασφαλής. Τι θα γίνει με αυτό το πρόβλημα, ο Σαλβάρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε από τον κύριο Ντεμέρα. είμαστε συνηθισμένοι να μας παραδίδει λεπτομερή και σωστή δουλειά και εδώ θα αναφερθώ ή στην τροπολογία του 8 γιατί ε, θα θέλαμε να υπάρξει μία διόρθωση παρόλο που βαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Ε, πρώτη φορά έρχομαι σε αυτή την Επιτροπή αλλά βλέπω ότι το θέμα αυτό δεν λειτουργεί και γι' αυτό ο εισηγητής έχει κάνει μία πρόταση. Ε, Παραδείγματο χάρη, η σχέση ε, και ρύθμιση Καναδά με την Τσεχική Δημοκρατία εφέτος. Ένα θέμα που έχει αναφερθεί από την κυρία Ρότοβα, ο κύριος Λαμπρινίδης και εγώ ο κύριος Ρίσκι και άλλοι είχαν προσυπογράψει διότι υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος δεν προωθεί έναν μια διμερή σχέση αλλά ένας μηχανισμός Ευρωπαϊκής Ενώσεως για πλήρη αλληλεπίδραση με τις τρίτες χώρες αφενός ένα θέμα το οποίο είχε ανα αναφερθεί ε, για το θέμα της Αυστρίας από τις Ηνωμένε Πολιτείε ότι θα επανέρχεται στις θεωρήσεις εάν δεν έδιδε τα, αυστρι... Ε, τα δακτυλικά αποτυπώματα οπότε φαντάζομαι ότι από αυτά σας προϋποθέσεις κάτι δεν πήγε καλά με τους εταίρους μας και δεν είναι δυνατόν να συνεργαστούμε έτσι με 27 κράτη-μέλη με τους συνεργάτες μας. Μετά ε, βλέπουμε το αρχικό κείμενο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, από το 2001 σχετικά με αυτό το θέμα. Οπότε υπήρχαν αυτόματοι μηχανισμοί αλληλεγγύης ε, και αλληλεπιδράσεως που προβλέποντο ε, και αν υπήρχε μία μείωση από ένα κράτος ίσχυε για όλα τα κράτη το 2001 για τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις. Τώρα όμως πολιτικά έχει βελτιωθεί η κατάσταση και γι' αυτό λέμε ότι βάσει της ε, ε, των τελευταίων εξελίξεων και τις προθεσμίες μας υπάρχει το περιθώριο των 90 ημερών και ο κύριος ε, Δίας Δεμέρα προτείνει να υπάρχει αυτομάτως υποβολή μίας προτάσεως αλλά εμείς προτείνουμε αυτό που έγινε στο Economic Governance Package δηλαδή να υπάρχει με ενισχυμένη πλειοψηφία που να χρησιμοποιηθεί και εδώ και μόνο εάν η ανισχυμένη πλειοψηφία των κρατών μελών αρνηθεί ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία ε, ε, απορρίψει την πρόταση αυτή ε, τότε να μην ισχύσει διαφορετικά η εφαρμογή να είναι αυτόματη για να υπάρχει μια ισορροπία και να δείξουμε στα κράτη-μέλη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει θεωρεί ότι είναι μία ένωση κρατών μελών που στηρίζονται όταν τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν προβλήματα από τρίτες χώρες και εάν συμφωνείτε με την ιδέα θα υποβάλουμε ε, την ε, τροπολογία αυτή γραπτός και επειδή υπάρχει μόνο μία τροπολογία δεν θα αναφερθώ στη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή τροπολογιών. Ο κύριος Ένσκου. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Δίας Δεμέρα για την εκθεσή του. Θα τον ευχαριστήσω και για το θάρρος του και την αλληλεγγύη που επιδεικνύει αναφέροντας στην έκθεση το ζήτημα του μηχανισμού αμοιβαιότητας. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα ήθελαν να ε, το αποφύγουν. Πιστεύω ότι αυτός ο μηχανισμός αμοιβαιότητας που προτείνεται αποτελεί σαφώς βελτίωση σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα συγκεκριμένο μέσο για την αμοιβαιότητα εκτός των διπλωματικών ε, διάβλων. οι διαπραγματεύσεις για τις θεωρήσεις μπορούν να διεξαχθούν μόνο από το Συμβούλιο και από την Κομισιόν και όχι από τα κράτη-μέλη. Η πρακτική μας έχει δείξει ότι τόσο η Κομισιόν όσο και το Συμβούλιο δεν ε, είναι ιδιαίτερα διατεθειμένα να υποστηρίξουν τα κράτη-μέλη όσον αφορά την αμοιβαιότητα των θεωρήσεων. Είναι σαφές ότι οι τρίτες χώρες ε, οι οποίες ε, δεν σέβονται την αρχή αμοιβαιότητα... θα πρέπει να καταλάβουν ότι έχουμε μια κοινή πολιτική για τις θεωρήσεις και ότι οι πολίτες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορούμε πλέον, δεν είναι δυνατόν πλέον η κοινή πολιτική για τις θεωρήσεις να οδηγεί σε, διακριτική, σε περίπτωση διακριτικής ε, μεταχείρισης. Πάνω από 100 εκατομμύρια ε, πολίτες είναι λιγότερο ίση από τους υπόλοιπα 400 εκατομμύρια. Έχω, ε, ήθελα να πω ότι η γραπτή δήλωση της κυρίας Ροϊφά δεν αφορά μόνο την Τσεχία αλλά και τις άλλες χώρες, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία και Κύπρο. Χώρες που δεν ε, απολαμβάνουν την αμοιβαιότητα για τις θεωρήσεις όσον αφορά τις σχέσεις τους με τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά. Μου κάνει έκπληξη ότι οι αντιπρόσωποι του Συμβουλίου και της Κομισιόν στις δηλώσεις τους δεν υποστήριξαν την ε, Ευρωπαϊκή Ενότητα. Αυτοί θα έπρεπε να είναι οι κύριοι υποστηρικτέ ε, της Ευρωπαϊκής Ένωση. Αυτοί θα έπρεπε να υποστηρίζουν κατά κύριο λόγο την Ευρωπαϊκή Ενότητα. Για ποιο λόγο πρέπει να γονατίζουμε μπροστά σε τρίτες χώρες. μας προβληματίζει το γεγονός ότι αντιμετωπίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον τρόπο στο πλαίσιο των διεθνών τη σχέσεων. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι αυτός ο μηχανισμός αμοιβαιότητας που παρουσίασε ο κύριος Ντεμέρα θα πρέπει να αναφέρεται καθαρά στις χώρες που ε, για τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν υποχρεώσεις ε, θεώρησης ε, για άλλα κρατημέλη. Υποστηρίζω αυτή την άποψη και θα υποβάλω μια τροπολογία για αυτό το ζήτημα. Ελπίζω ότι τα μέλη θα με υποστηρίξουν, διότι, όπως φαίνεται εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαστε οι μόνοι που θέλουμε αυτή την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κυρία Ρόιτοβα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας και τον κύριο Άλβαρο που αντελήφθηκαν με πόσο επίκαιρο είναι το θέμα της αμοιβαιότητας για την ενότητα των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και τέσσερις μήνες περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εκπροσωπεύει τα συμφέροντα των χωρών μελών σε ό,τι αφορά την αμοιβαιότητα για θέματα θεωρήσεων. Και ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή που συμπεριέλαβε τη σχετική τροπολογία. Θα πρέπει να διατρανώσουμε την επιθυμία μας να εμείνουμε στις θέσεις μας και να μην υπαναχωρήσουμε. Και είναι σημαντικό και το Συμβούλιο, από ό,τι φαίνεται, τα λεγόμενα της Πολωνικής Προεδρίας αντιλαμβάνεται το διακύβευμα εδώ. Υπάρχουν ε, ακραίες καταστάσεις όπως μεταξύ Καναδά και Τσεχίας, αλλά δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε στο διμερές επίπεδο για να επιλύουμε τα σοβαρά αυτά προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των κρατών μελών. Φαίνεται όμως ότι αδιαφορεί γι' αυτό. Αδιαφορούν επίτροποι και αδρανούν, δεν δραστηριοποιούνται για την ενεργό προάσπιση των συμφερόντων μας. Και δεν είναι μόνο ε, πρόβλημα ο Καναδάς, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Για παράδειγμα, τι γίνεται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ε, για τις παλιές χώρες μέλη ισχύει υποχρέωση, ισχύει απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης. Οι νέες όμως χώρες, οι υπήκοοι των νέων χωρών έχουν υποχρέωση θεώρησης για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Γιατί να μιλήσουμε αυτό το πρόβλημα με την παράγραφο 10. Προσπαθούμε να βρούμε λύση. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδρά στη δήλωση που ενέκρινε η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει κάτι εδώ που δεν λειτουργεί σωστά. Υπάρχει κι άλλο σοβαρό πρόβλημα. Οι Τσέχοι πολίτε όταν ζητούν βίζα χρειάζεται να περιμένουν τρεις με πέντε εβδομάδες και πολλέ φορέ χρειάζεται να πάνε και δύο φορές ε, στην Πράγα με τα συναφή έξοδα για να συμπληρωθούν ε, βέβαια τα αποσπάσματα τραπεζικών λογαριασμών και ε, οι διατυπώσεις που πρέπει να περάσουν οι Τσέχοι πολίτες για να πάρουν βίζα για τον Καναδά είναι δυσβάσταχτες. Επίσης το θέμα της υιοθεσία αναφέρεται. Και μερικές φορές στρέφονται οι Τσέχοι πολίτες σε μένα και μου λένε ε, παραβιάζουν κάποιο κανόνα. Δεν θεωρούν ότι ε, χορηγία προς ένα εξαποστάσεως σε ένα παιδί του τρίτου κόσμου θα πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά ε, στο έγγραφο για την αίτηση ε, βίζας. Γιατί δεν ε, ισοδυναμεί με υιοθεσία μια τέτοια κατάσταση. Γιατί λοιπόν ο Καναδάς απαιτεί και τέτοιες περιπτώσεις να αναφέρονται στις διατυπώσεις. Νομίζω ότι έτσι δημιουργούνται μεγάλα χάσματα μεταξύ ημών και των ευρωσκεπτικιστών, με τέτοιες υποθέσεις που ουσιαστικά ρίχνουν νερό στο μήλο των ευρωσκεπτικιστών. Επανερχόμαστε στον εισηγητή μα, τον κύριο Δία Δεμέρα, για να απαντήσει στα σχόλια. Α, συγγνώμη κύριε Μπρόγκ, ε, δεν σα πρόσεξα. Θα ακούσουμε πρώτα εσά και μετά τον κύριο Δία Δεμέρα με το να αφαιρέσουμε την ανάγκη ε, ε, για τις θεωρήσεις εσείς ξεκινάτε από την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει αύξηση της παράνομης ε, μετανάστευσης πράγμα το οποίο είναι κάτι θετικό αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μία αύξηση των μετακινήσεων και δεν πιστεύουμε ότι αυτό θα λειτουργήσει ακόμη και υπό προϋποθέσεις υπάρχουν χώρες με χαμηλότερο κατακεφαλή είναι εισόδημα, ανεπαρκείς υποδομές, κακές κοινωνικές υπηρεσίες, κάποιο επίπεδο μετανάστευσης είναι αναπόφευκτο και περισσότερο στην Ευρώπη από ότι οπουδήποτε αλλού για προφανείς λόγους. Υπάρχει λοιπόν μία διαφοροποίηση μεταξύ των νομίμων επισκεπτών και των παρανόμων για την Αυστραλία είναι πολύ εύκολο να αποκτήσει κανείς θεώρηση ηλεκτρονικά όπως εγώ όταν την επισκέφτηκα. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε ε, να αφαιρεθεί η ε, ε, απέτηση θεώρησης όταν υπάρχει η δυνατότητα παράνομης με τα κίνησης αλλά πιστεύω ότι ε, ε, αν υπάρχει η θεώρηση είναι πολύ μικρότερος ο κίνδυνος να παραμείνει κανείς περαιστέρω από ό,τι διαφορετικά και τώρα ο εισηγητής Δίας Δεμέρα έχει το λόγο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Νομίζω ότι το πρώτο συμπέρασμα από τη συζήτηση είναι ότι δεν έχουμε ένα μικρό τεχνικό ζήτημα. Είναι με τεχνικό το θέμα, αλλά έχει τεράστιο πολιτικό αντίκτυπο. Ε, θα δώσω τώρα κάποιες απλές εξηγήσεις. Θα έχουμε άλλη ευκαιρία για πιο διεξοδική ανάλυση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως για τα σχόλια που έκανε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει με θετικό μάτι και την έκθεση και τις τροπολογίες. Θεωρεί ότι οι τροπολογίες βελτιώνουν την πρόταση και ε, υπέβαλε κάποιες επιφυλάξεις ως προς τη θέση του εισηγητού για το μηχανισμό της αμοιβαιότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με την εξαίρεση ε, για ε, τις θεωρήσεις για τα μέλη των πληρωμάτων ότι αφορά την τροπολογία 11 που είναι η τροπολογία της αναστολής, του μηχανισμού αναστολής, θα ήθελα να διευκρινίσω και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά να εξηγήσω και στους συναδέλφους που είχαν την απορία ότι η τροπολογία αυτή σε καμία περίπτωση δεν θέλει να καταστρατηγήσει τη νομική βάση της επιτροπολογίας, το σχετικό άρθρο που αποτελεί τη βάση της ε, επιτροπολογίας. Σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει πρότασή μου το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το αντίθετο, αυτό που επιδιώκουμε και το επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω εδώ, αυτό που επιδιώκουμε... Ε, εκφράζοντας την βούληση που έδειξε και ατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό μας ενδιαφέρει. Η παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όχι μόνο από τη στιγμή έναρξης της διαδικασίας, αλλά από την στιγμή που ένα κρατος λαμβάνει γνώση της υπόθεσης αυτής, από προηγούμενο δηλαδή στάδιο, σε ό,τι αφορά τα μαθηματικά κριτήρια τα αριθμητικά, μαθηματικά κριτήρια. Προσπαθώ εδώ να απαντήσω στις ερωτήσεις που έγιναν για τα ποσοστά. Τα μαθηματικά αυτά τα αριθμητικά κριτήρια έχουν στόχο να αποφύγουν την αυτόματη εφαρμογή του μηχανισμού και να δημιουργήσουν μια ελαστικότητα. Τώρα τα μαθηματικά αριθμητικά κριτήρια 50%, 60% αυτό είναι υποδιαπραγμάτευση θέμα, είναι συζητήσιμο, δεν είναι κάτι άκαμπτο και είναι και η αφετηρία, όπως είπα προηγουμένως. Συμφωνώ πάντως ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Η αμοιβαιότητα, κατά τη γνώμη μου, εξηγείται με διεξοδικό τρόπο στην τροπολογία 10. Στόχος της πρότασης αυτής είναι η ελαστικότητα, η μεγαλύτερη ελαστικότητα. Και θα ήθελα και πάλι να καθησυχάσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εισηγητής είναι πρόθυμος για διαβουλεύσεις και συζήτηση. Σε καμία περίπτωση στόχος της πρότασης του συγητού δεν είναι η παραβίαση οποιασδήποτε συνθήκη ή οποιαδήποτε διάταξη. Αυτό που διεκδικούμε είναι η παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλε τι φάσει τη διαδικασία. Από τι πρώτερε φάσει. Σε ορισμένε φάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να είναι ω απλό προσκεκλημένο, σε άλλε φάσει με βάση τη διαδικασία συναπόφαση ω πλήρε μέλο τη διαδικασία αυτή. Επαναλαμβάνω, αυτό το δικαι... αυτή η πρόταση του εισηγητού συνάδει πλήρως με το δικαίωμα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σεβόμαστε απόλυτα τους κανόνες της τροπολογίας. Αυτή είναι η απάντησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, θα ήθελα να εκφέρω την απόλυτη μου διάθεση και προθυμία για την ε, ανέβρεση λύσεων. Κύριε Φιλίπ Ζαριζισκή, εκπρόσωπε του Συμβουλίου. Θα ήθελα να εκφράσω την ε, βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου προς την Πολωνική Προεδρία και προσωπικά προς τον κύριο Ζαζίνσκι για την ε, μεγάλη προθυμία του και το πνεύμα συνεργασία που έδειξε καθ' όλη τη διάρκεια των συζητήσεων. Συμφωνώ ότι αυτό το θέμα είναι το μείζον ζήτημα τη ομάδα εργασία του Συμβουλίου για τι Θεωρήσει. Ξέρω ότι ε, δόθηκαν πολλέ πληροφορίε και έγινε πολύ διεξοδική ενημέρωση και αν η ομάδα εργασία για τις θεωρίες θέλει ισορροπία, αυτό είναι το ζητούμενο και για τον εισηγητή. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε στενέ επαφέ μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο και ο εισηγητή, ο υποφαινόμενο και οι σκιώδει εισηγητέ. Κάτι άλλο που είπαν πολλοί συνάδελφοι είναι ότι τα δύο ουσιώδη ζητήματα της έκθεση αυτή είναι η ρήτρα διασφάλιση και η ρήτρα αναστολή. Θα πρέπει να λειτουργήσουν και τα δύο θέματα. Αν δεν καταφέρουμε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά αυτά τα δύο ζητήματα, δεν έχει νόημα το έργο που κάνουμε. Θα πρέπει να αποφύγουμε τη διακριτική μεταχείριση. Σε ό,τι αφορά την αναστολή, μερικοί είναι υπέρ τη διατήρηση των ποσοστών. Εγώ όχι. Εγώ είμαι υπέρ τη διαπραγμάτευση για τα ποσοστά. Τα ποσοστά είναι ένα εργαλείο, είναι ένα μέσο για να αποφύγουμε οποιαδήποτε αυτοματισμό στην εφαρμογή του μηχανισμού κάθε ε, περίπτωση αναστολής θα πρέπει να εξετάζεται με μεγεθυντικό φακό, διεξοδικότητα και περιπτωσιολογικά και τα ποσοστά είναι ένα επιπλέον στοιχείο, αλλά δεν είναι το αποφασιστικό στοιχείο στην ε, εξέταση ενός φακέλου. Επίσης θα πρέπει να αξιολογήσουμε στη διαδικασία και την έκθεση της Frontex, ε, της Europol, της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Γραφείου για το Άσυλο και να λάβουμε υπόψη και τη, θε, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Μερικοί συνάδελφοι και ο κύριος Νατζίνσκι αναφέρθηκε σε αυτό ότι άλλος ο αντίκτυπος στη Γερμανία και άλλος ο αντίκτυπος στο Λουξεμβούργο Συμφωνώ απόλυτα. Άσχετα λοιπόν με το γενικό θέμα, και εδώ θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Άλβαρο, σίγουρα στη, στα θέματα αμοιβαιότητας καλύτερα να έχουμε συνεργασία 27 χώρες μέλη και να μην α, α, υιοθετούμε κατακαιρματισμένη προσέγγιση και έχουμε κατά περίπτωση μόνο συζήτηση. Η αλληλεγγύη είναι επίση απαραίτητη. Γι' αυτό και θέλουμε συνεργασία σε επίπεδο 27 χωρών μελών, αλλά η ανάλυση γίνεται περιπτωσιολογικά και όλα τα υπόλοιπα είναι εργαλεία για να ε, αξιολογήσουμε το κατά πόσο θα λάβει η χώρα τελικά η αναστολή από την υποχρέωση απαλλαγής. Επαναλαμβάνω πάντως ότι έχουμε κάποια μαθηματικά στοιχεία, δεν είναι ο απόλυτος κανόνας. Όλοι θέλουμε συνένεση. Αυτό είναι το ζητούμενο, να καταλήξουμε σε συμφωνία. Και τέλος, συνάδελφοι, νομίζω ότι στείλαμε ένα χειρό μήνυμα προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα αυτό δεν είναι μόνο θέμα του εισηγητού. Το θέμα αυτό είναι κοινό. Είναι μέλημα όλων υπάρχει ευρεία συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορούμε να το πούμε αυτό χωρίς ματαιοδοξία, με ταπεινοφροσύνη αλλά με ρεαλισμό, υπάρχει ευρεία συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως εκφράστηκε από τη συζήτηση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Αυτή η συνένεση είναι πολύ σημαντική για τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Φαγιόν, συμφωνώ με αν συμφωνούν και οι υπόλοιποι, αν προτιμάτε την 6η Δεκεμβρίου 12 το μεσημέρι ω καταληκτική διορία για την υποβολή τροπολογιών, δεν έχω αντίρρηση. 6 Δεκεμβρίου 12 το μεσημέρι. Συμφωνώ και εγώ ότι ο μηχανισμός αναστολής είναι καλύτερη διατύπωση και σας ευχαριστώ που συμφωνείτε με την πρότασή μου και ευχαριστώ Τάνια που προτείνεται ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Χωρί όμω καταστρατήγηση τη διαδικασία τη επιτροπολογία αλλά απλώ δίνοντα το παρόν ω προσκεκλημένη στην Επιτροπολογία. Σε ό,τι αφορά την αμοιβαιότητα, ευχαριστώ πάλι την Σκιώδη Συγγήτρια που τάχθηκε υπέρ του μηχανισμού, γιατί ο μηχανισμό αυτό συνάδει και με τη ελληνική. <clears throat> Και με το ψήφισμά μας του Μαρτίου του 2011, το οποίο συζητήσαμε και υπογράψαμε. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ζήτησε κατάργηση των ποσοστών. Εγώ σας είπα τι, ποια είναι η γνώμη μου. Είναι ζήτημα διαπραγμάτευση τα ποσοστά. Να αποφύγουμε πάση θυσία τον αυτοματισμό. Γι' αυτό υπάρχουν τα ποσοστά, αλλά δεν είναι το αποφασιστικό κριτήριο. Ε, ευχαριστώ, Τάνια, για την ε, ε υποστήριξη των τροπολογιών και τη δήλωση ότι δεν θα υποβάλει στι δικέ τροπολογίε. Ευχαριστώ και τους, ε, την, ε, ε, συντονίστρια τη Άλντε για τα θετικά σχόλια, τα ανταποδίδω. Όντω η έκθεση αυτή έχει και ένα τεχνικό σχέλο, αλλά και ένα πολιτικό σκέλος. Και συμφωνώ με τη Ρένατε Βέμπερ ότι ανάγκη ε, έχουμε για κατοχύρωση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Γιατί η αλληλεγγύη βρίσκεται στα γονίδια μας. Στα γονίδια και τα δικά μας ως πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στα ίδια τα γονίδια της συνθήκης Λισαβόνας. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σου, Ρενάτε. Έκανες δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τα ποσοστά, το 50% και το 60% για τα ποσοστά μίλησα. Τα ποσοστά υπάρχουν για να μην εφαρμόζεται αυτόματα ο μηχανισμός. Για να υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα και δυνατότητα περιπτωσιολογικής ανάλυσης της κάθε περίπτωσης. Επειδή είσαι και νομομαθής, φυσικά ενδιαφέρεσαι για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στη διαδικασία τη επιτροπολογία. Είσαι και καλή νομικό, δεν χρειάζεται να ανησυχεί καθόλου. Σε καθησυχάζω, γιατί αν διαβάσει με προσοχή την τροπολογία μου, θα διαπιστώσει ότι σε καμία περίπτωση η πρόταση αυτή δεν καταστρατηγεί τη διαδικασία τη επιτροπολογία. Θέλουμε απλώ το Κοινοβούλιο να προσκαλείται στη διαδικασία αυτή, ακολουθώντα φυσικά συστάσει τη ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητούμε πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν την επίσημη έναρξη τη διαδικασία. Κύριε Μπουσούτιλ, ευχαριστώ Σάιμον. Ευχαριστώ για την πραγματικά έθεση των δάκτυλων επί των τύπων των ύλων. Όντω θέλουμε ένα σύστημα θεωρήσεων που θα είναι αξιόπιστο. Και για να είναι αξιόπιστο αυτό το καθεστώ των θεωρήσεων, χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό αναστολή που θα λειτουργεί αποτελεσματικά. Το είπε με μεγάλη ακρίβεια και πολύ σωστά. Και σε ευχαριστώ θερμά. Δύο διευκρινήσει ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα και την περίπτωση κατάχρηση δεν θέλω να μακρηγορήσω, σε παραπέμπω στην τροπολογία 10 και στην τροπολογία 11. Ε, και επίσης, Σάιμον, απάντησα και για τις καταχρήσεις και για το διαφορετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν σε μια χώρα που έχει τις διαστάσεις του Λουξεμβούργου ή μια χώρα που έχει τις διαστάσεις της Γερμανίας, της Σλοβενίας ή της Ισπανίας. Κυρία Ζήπελ, όπως γνωρίζετε κι εσείς, υπάρχει ένας θετικός κατάλογος και ένας αρνητικός κατάλογος. Το παράρτημα 1 και το παράρτημα 2 δηλαδή. Αλλά δεν είναι απεριορίστου διαρκείας. Από το 2001 που τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός έχει τροποποιηθεί 8 φορές. Βρίσκεται σε μία διαδικασία συνεχούς αναθεώρησης ε, και μεταμόρφωσης αυτός ο κανονισμός. Ανάλογα με τις διάφορες καταστάσεις που ανακύπτουν μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών που βρίσκονται στον πρώτο κατάλογο ή στο δεύτερο, στο πρώτο παράρτημα ή στο δεύτερο. Κύριε Άλβαρο, ευχαριστώ Αλεξάνδερ για τα λόγια σου και την συμφωνία σου με την τροπολογία 10. Σε ό,τι αφορά την αμοιβαιότητα, συμφωνώ και εγώ ότι ο μηχανισμός δεν λειτουργεί και γι' αυτό έχει νόημα να υποβάλουμε μια πρόταση αναθεώρησης. Αναφερθήκατε στην περίπτωση του Καναδά. Και εσείς Άλβαρο και εγώ συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε έναν κοινοτικό κανονισμό. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο κοινοτικό κανονισμό όχι μόνο για να είμαστε αλληλέγγυοι, αλλά για να έχουμε και αξιοπιστία. Και είδαμε τη διαστρεβλωτικά αποτελέσματα έχουν οι απαιτήσει για τα δακτυλικά αποτυπώματα μεταξύ ΗΠΑ και Αυστρίας. Το 2001 είχαμε αυτόματη αμοιβαιότητα. Τώρα προτείνεται οι 90 ημέρες. Περιμένω την τροπολογία σας, κύριε Άλβερο. Θα την συζητήσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Κύριε Έντσιου, ευχαριστώ θερμά αγαπητοί συνάδελφοι για τα σχόλιά σου. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας, ε, κυρίως για το σχόλιο ότι με την έκθεση βελτιώνεται ο μηχανισμός αμοιβαιότητας. Συμφωνώ ότι ένα μηχανισμό θεωρήσεων, ένα σύστημα θεωρήσεων, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δημιουργεί διακριτική μεταχείριση μεταξύ των 27 χωρών μελών. Περιμένω και τη δική σα τροπολογία. Θα την εξετάσουμε προκειμένου να εντοπίσουμε και άλλες χώρες όπως η Ρουμανία πέραν της Τσεχίας που πλήττονται από αυτή τη διακριτική μεταχείριση που εμείς θέλουμε πάση θυσία να αποφύγουμε. Κυρία Ρόιτοβα, σας ευχαριστώ και σας για τα σχόλιά σας και τη συμφωνία σας με την θέση του κυρίου Άλβαρο. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα των χωρών μελών. Προσπαθεί όμως, προσπαθεί να μας εκπροσωπήσει όλους. Καταβάλει τετάνιες προσπάθειες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταλήξει σε συμφωνίες και συνενετικές λύσεις, όπως και στην περίπτωση αυτή. Και συμφωνώ μαζί σας ότι η δική μας πρόταση για την αμοιβαιότητα, η δικιά σας και η δικιά μου, δεν είναι για πέταμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της. Μίλησατε για την περίπτωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και είπατε ότι κρίμα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντέδρασε κατεπηγόντως σε περιπτώσεις ε, διαφοράς όπως αυτή που ανέκυψε μεταξύ Καναδά και Τσεχίας. Επίσης, ε, είπατε ότι είναι και καινή ώρα για δράση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας κυρία Ρότοβα. Ο κύριος Μπρόγκς εξέφρασε ανησυχίες ό,τι αφορά το μηχανισμό της αναστολής και είπε ότι κατά τη γνώμη του η αμοιβαιότητα είναι άσχετο θέμα με την υπόθεση αυτή. Δεν συμφωνώ κύριε Μπρόγκς με την ε, διαπίστωσή σας ότι η αμοιβαιότητα εδώ είναι άσχετο ζήτημα. Το αντίθετο είναι πολύ σημαντική και μάλιστα με το ψήφισμά μας του Μαρτίου του 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε την αμοιβαιότητα ως σημαντικό δόγμα γιατί έχουμε αμοιβαιότητα ή ε, 27 και ε, περιπτωσιολογική αμοιβαιότητα. Κύριε Πρόεδρε, αφιερώσαμε πολύ χρόνο, αλλά το θέμα είναι πραγματικά σημαντικό. Σας ευχαριστώ όλους για την καλή σας θέληση και ευχαριστώ το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω να τα λάβουν όλα αυτά υπόψη με ταπεινοφροσύνη, αλλά παρόλα αυτά να λάβουν υπόψη την κοινή αυτή θέση που πραγματικά είναι κοινή και συνενετική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Δίας Δεμέρα. Είχαμε ευρεία συζήτηση, μακροσκελή, εξετάζοντας το σχέδιο έκθεσης και από ό,τι κατάλαβα συμφωνήσαμε ως διορία για την υποβολή τροπολογιών την 6η Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Συμφωνεί και ο εισηγητής, 6 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι λίγη προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, όπως πρότεινε η η κυρία Τάνια Φαγιών. Περνάμε στο επόμενο θέμα με ολιγόλεπτη καθυστέρηση, γι' αυτό και καλό θα ήταν να, να κερδίσουμε αυτό το χαμένο χρόνο. Μια και το επόμενο θέμα μετά την έκθεση που θα συζητήσουμε είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Γι' αυτό καλό θα ήταν να μην καθυστερήσουμε και να μην ξεχάσετε και τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας παρακαλώ. Το επόμενο θέμα λοιπόν είναι η τροποποίηση του κανονισμού που θεσπίζει κοινοτικό κώδικα θεωρήσεων. Η συγητής μας για το θέμα αυτό είναι ο κύριος Λουί Μισελ που θα μας κάνει και την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης του. Κατόπιν θα ακούσουμε εν συντομία, και το τονίζω, εν συντομία, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον εκπρόσωπο της Πολωνικής Προεδρίας. Κύριε Λούιμισέλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να μπορέσω να σας κερδίσω χρόνο σε σχέση με την ημερήσια διάταξη, διότι όπως ελέγχθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, προσπαθούμε τεχνικά να βελτιώσουμε τις διατάξεις που αναφέρονται εις εις θεωρήσεις διέλευσης από αεροδρόμιο, διότι λέγεται ότι όσοι έχουν αδία παραμονής ή η ε, νόμιμη θεώρηση σε χώρα που δεν εφαρμόζει το σύστημα Σένιεν όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και άλλες ε, μπορούν να έχουν μία θεώρηση για διέλευση από το αεροδρόμιο. Δεν αλλάζουμε δηλαδή τις πρακτικές των κρατών μελών στην παρουσίαση της, ε, του θέματος στην Επιτροπή αυτό δεν έθεσε προβλήματα γι' αυτό και στηρίζω την πρόταση και ζητώ από την Επιτροπή Ελευθεριών να ε, ε, στηρίξει την πρόταση αυτή με δύο τροπολογίες ή στα εκτιμώντας 10 και 11. Αυτό είναι όλο κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μέσα στην αίθουσα. Ωραία, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την σύντομη παρουσίαση της εκθέσεώς του που αντικατορπτρίζει ακριβώς τη συμφωνία που επετεύθη στην παρουσία και την πρώτη συζήτηση στην Επιτροπή Ελευθεριών ε, για τα ε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει τα, ε, τις δύο τροπολογίες διότι συνάδουν με τις τροπολογίες οι οποίες υιοθετήθηκαν στο Συμβούλιο. Τώρα εκπρόσωπος της Πολωνικής Αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς συμφωνούμε πλήρως, είναι εξαιρετική κατάσταση, βλέπουμε ότι τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται στενά και είμαστε ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ. Και αυτό ήταν πολύ σύντομο. Η κυρία Ζόμερ έχει ζητήσει το λόγο και της τον δίδω και εγώ μία σύντομη παρατήρηση. Συμφωνώ με τον εισηγητή, δηλαδή νομίζω ότι αυτή η τεχνική προσαρμογή είναι σωστή και αυτό απεδείχθηκε στη χρήση. Ότι δηλαδή υπάρχει ακόμη ένα λιθαράκι για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί το οικοδόμημα και ευχαριστώ τον εισηγητή και πιστεύω ότι το ΕΛΚΑ θα τον στηρίξει. Ευχαριστώ και πάλι. Ο κύριος Ενσού. Ε, ευχαριστώ. Σαν εισηγητής ε, της ε, ε, Επιτροπής στηρίζω τον σαν σκιώδη εισηγητή στηρίζω αυτή την έκθεση και πιστεύω ότι δεδομένη της τεχνικής μορφής δεν χρειάζεται πολλά σχόλια. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι ε, είναι το καλύτερο ε, για την Ρουμανία και τη Βουλγαρία να υιοθετηθούν ή στην ε, ζώνη Σένιαν, οπότε δεν θα χρειάζονται τέτοιες τροπολογίες. Ευχαριστώ διότι έτσι καλύψαμε το χρόνο και μπορούμε να επανέλθουμε στον κύριο Μισελ αν θέλει να κλείσει τη συζήτηση αυτή χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε λοιπόν για αυτό το θέμα. Και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες όπως έχουμε προτείνει και θα ψηφίσουμε. Εδώ Έχουμε στο σημείο 7 την κατάρτιση ενός μηχανισμού αξιολογήσεως για να επαληθεύεται η εφαρισμογή ε, του κεκτημένου Σένιεν που είναι ε, η έκθεση του συναδέλφου Κάρλος Κοέγιο και υπάρχουν ορισμένες συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες έχουν υποβληθεί στον εισηγητή και ο εισηγητής ε, είναι έτοιμος να στηρίξει την έκβαση των ε, διαπραγματεύσεων και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόκειται να έχουμε μία φοφορία προσανατολισμού το αποτέλεσμα του συμβεβασμού μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Και ήθελα να υπογραμμίσω τέσσερα σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω ε, για την καλή συνεργασία με τους κοιόδους και την μεγάλη συνένεση που επετεύχθη στην Επιτροπή μας, τη ΛΥΜΠΕ. Στο δεύτερο σημείο θέλω να υπογραμμίσω ότι πραγματικά χρειαζόμαστε ένα πραγματικό μηχανισμό αξιολόγησης του χώρου Σέγγεν. Η ασφάλεια του χώρου Σέγγεν βασίζεται στην δίκαιη και αποτελεσματική αξιολόγηση. Το τρίτο πράγμα που ήθελα να πω είναι ότι προσπάθησα να αποδεχθώ τις περισσότερες τροπολογίες των υπολοιπών συναδέλφων. Ωστόσο, ορισμένες από αυτές δεν μπορούσα να τις δεχθώ λόγω της διαίρεση του αρχείου σε δύο διαφορετικές προτάσεις και λόγω νομικών περιορισμών. Το, η τέταρτη μου και τελευταία παρατήρηση είναι ότι θέλω να πω ότι με αυτή την ψηφοφορία ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διατεθειμένο να εξετάσει μαζί με το Συμβούλιο και την Κομισιόν οποιασδήποτε δυνατές νομικές λύσεις που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε συμβιβασμό μεταξύ των τριών οργάνων. Πιστεύω ότι, κυρία Πρόεδρε, είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ε, θα ε, κάνουμε μια ψηφοφορία ενδεικτική ψηφοφορία και βάσει του αποτελέσματος θα ξεκινήσει ο συγκητής της διαβουλεύσεις με τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ξεκινάμε όλοι έτοιμοι, κυρία Μέγκστρομ. Δεν φέρετε την ηλεκτρονική σας κάρτα. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Ζητώ συγγνώμη, δεν έβρισκα την κάρτα ψηφοφορία μου. Μπορείτε ωστόσο να λαμβάνετε υπόψη την ψήφο μου ούτω ή άλλω. Ευχαριστώ. Ναι, εντάξει. Δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Είναι η πρώτη φορά. Συμβαίνει, συμβαίνει και στους καλύτερους. Ναι κύριε Τριανταφυλλίδη και το ίδιο και εγώ παρακαλώ. Μάλιστα, ξεκινάμε. Έχετε όλη την λίστα συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μία αποχή. Ορισμένες καταπίπτουν και περνάμε στην προφορική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην προφορική τροπολογία 2. Τροπολογία, συγγνώμη, 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε τώρα στη συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 υπέρ κατά κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική 4 όχι προφορική 4 υπέρ κατά κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές θα το ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 64 άρχεται η ψηφοφορία Κλείνει η ψηφοφορία. Δεν μπόρεσα να ψηφίσω. Λέει κάποιο με την κάρτα. Δεν έχω την κάρτα ψηφοφορίας μου, αλλά ψηφίζω κατά. Μπορείτε να καταχωρήσετε την ε, ψήφο μου κατά, παρότι δεν μπορώ να ψηφίσω. Εσείς ψηφίσατε υπέρ. Και ο κύριος Τρενταφυλίδης Ωραία, θα ξαναελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Η κάρτα μου τώρα λειτουργεί. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ψηφίζετε. Κλείνει η ψηφοφορία. Τι έχουμε. Κύριος Τρενταφυλίδης είναι υπέρ. Ε, έχω τώρα την κάρτα μου ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Πόρο η Βίξτρομ λοιπόν. Υπέρ. Και εγώ ψηφίζω κατά, λέει ο κυρίος. 21 με 23 και εγκρίνεται. ...23 υπέρ και 22 κατά. Ωραία, την ξανακάνουμε, την ψηφοφορία. Κυρία Βίξτρομ, εσείς ψηφίζετε υπέρ, χωρίς κάρτα. Με δύο επιπλέον κατά και ένα υπέρ εγκρίνεται, αλλά μπορούμε να ξαναελέγξουμε αν θέλετε. Το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ξαναψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Βίξτρομ ψηφίζει υπέρ 23 εναντίον 22 εγκρίνεται εγκρίνεται περνάμε στην προφορική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία ε, ε συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 αποσύρεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές ε, ελέγχουμε για την 71 Ψηφίζουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία. 71 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 72 με υπάρχει μια προφορική τροπολογία εδώ από ό,τι κατάλαβα το representative 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται νομίζω περνάμε στην συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και προφορική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τα εκτιμώντας τώρα συμβαστική 11 στο πρώτο εκτιμώντας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 τώρα περνάμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε σε 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ορισμένες καταπίπτουν περνάμε στην προφορική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα ψηφίζουμε το κείμενο τελική ψηφοφορία όπως έχει τροποποιηθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Βίξτρομ, μία επιπλέον ψήφος υπέρ, το οποίο σημαίνει 42 υπέρ, καμία κατά, καμία αποχή, τέσσερις αποχές, 43 υπέρ λοιπόν, συγχαρητήρια κύριε Κοέλιο. Και τώρα αυτό σημαίνει ότι περνάμε στο σημείο 8. Παρουσίαση των προτάσεων της Επιτροπής. Θα ακούσουμε μια παρουσίαση από τον κύριο Στέφανο Μανσερβίση, Γενικό Διευθυντή της ε, Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων του χαρτοφυλακίου εσωτερικών υποθέσεων ωστόσο δεν βρίσκεται ακόμη εδώ για να κάνει την παρουσίαση του σχετικά με τα χρηματοδοτικά προγράμματα στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων για τα επόμενα ε, χρόνια. Προτείνω λοιπόν να κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα ώστε να μπορέσει να, να τον περιμένουμε. Σε 10 λεπτά συνεχίζουμε. Ευχαριστώ.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

Bueno,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

Ευχαριστώ.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 Ναι. Ναι, λοιπόν, είπαμε διάλειμμα ως 11.30, αλλά τώρα είναι 11.30. Οπότε, αν είναι ε, ήδη είναι ακόμη έξω, καλά θα είναι να έρθουν. Οπότε έχουμε μία ώρα μπροστά μας, ήταν το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Λοιπόν, ε, ξεκινάν και πάλι οι εργασίες μας. Είχαμε ένα διάλειμμα 10 λεπτών ε, περιμένοντας ε, τον κύριο Μαντσερβίση να έρθει. Είναι εδώ ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικών Υποθέσεων ο οποίος θα μας παρουσιάσει την νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία των δύο ταμείων ε, ε, στον ε, τομέα των εσωτερικών υποθέσεων από το 2014 έως το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει αυτές τις προτάσεις και δίνουμε το λόγο στον κύριο Μασεβίση ο οποίος θα μας παρουσιάσει τις προτάσεις αυτές και μετά θα γίνει συζήτηση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και πάλι για την, ε, ε, ε, την πρόσκληση να έρθω εδώ να παρουσιάσω εδώ την χρηματοδότηση στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο των εσωτερικών υποθέσεων. Ήδη το Μάρτιο είχα παρουσιάσει τις θέσεις μας και τους προσανατολισμούς μας και όπως είπατε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει την ανακοίνωση του Ιουνίου για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και 15 Νοεμβρίου όπως είπατε συμπληρώσαμε επίσης το πρόγραμμα και το πακέτο με την νομοθετική και νομική βάση. Ουσιαστικά αυτό που σας είπα <clears throat> ήταν ότι η πρόταση την οποία προτείναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε αποδεκτή και τώρα έχουμε προτείνει κάτι το οποίο πρόσχεται πολύ στις αρχιτικές μας ιδέες από πλευράς χρηματοδότησης και χρήσεως των πόρων αυτών στο μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω <clears throat> και να σας υπενθυμίσω καταρχήν ότι... Ε, κοιτάζοντας την χρηματοδότησή μας πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη δύο στοιχεία. Καταρχήν ότι στο προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στην ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε η απέτηση να γίνουν περισσότερα, γρηγορότερα, περισσότερα αναλογικά διότι οι εσωτερικές υποθέσεις είναι στο επίκεντρο του παντός και η διαχείριση αυτή ε, μέσα στο χρόνο πρέπει να αυξάνεται, πρέπει ε, να αντιληφθούμε ότι έχουμε συνεχώς νέες πιέσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίζουμε και άρα ε, ένα σημείο αναφοράς ήταν η αύξηση της ζητήσεως, δεύτερον η χρησιμοποίηση και αξιολόγηση των διαθεσίμων πόρων, όχι μόνο για να δούμε αν χρειαζόμαστε περισσότερα, αλλά για να δούμε <clears throat> πώς μπορούσαμε να επιτύχουμε τους στόχους των πολιτικών τους οποίους επιζητούσαμε και εδώ προσωπικά όταν ήρθα και εδώ ήταν ότι έπρεπε να ενισχύσουμε τα μέσα που διαθέταμε τα οποία ίσως δεν ήταν τόσο προφανή δεύτερον ότι ε, οι προκλήσεις διοικητικά ήταν τεράστιες και γι' αυτό ε, κάθε χρόνο έπρεπε να υιοθετούμε πέραν των 100 αποφάσεων για τα κράτη-μέλη, για τα προγράμματα εργασίας και ε, πέραν του ότι ήταν κάτι το επίγον έπρεπε να μετακινηθούν ε, χρήματα από τον ένα τομέα στον άλλον που πολλές φορές δεν ήταν αναγνωρίσιμα και προσέθεταν γραφειοκρατικό βάρος και αυτό θεωρήσαμε στην αρχή σαν το κρίσιμο σημείο και η κρίσιμη εμπειρία που είχαμε βιώσει και γι' αυτό τώρα έχει υιοθετηθεί το πρόγραμμα το οποίο επιτρέπει να υπάρξει μία αρχιτεκτονική η οποία είναι απλοποιημένη και είναι πολύ πιο άμεση σε σχέση με τους στόχους δηλαδή ε, έχουμε τώρα αντί για διάφορα ταμεία, δύο ταμεία, ένα για την ε, μετακίνηση και ε, τη διαχείριση των συνόρων και ένα για το άσυλο και, τη, και ε, έτσι καλυπτόμεθα από τις συνθήκες. Δεύτερον, έχουμε τονίσει την τεχνική κοινή διαχείρισης, δηλαδή αναδιαρθρώνουμε τον το τομέα που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι τώρα υπάρχει κοινή διαχείριση και των δύο τομείων και πλέον και της ασφαλείας που μπορούμε να στηρίξουμε ορισμένα προγράμματα και υπάρχει αυτή η κοινή διαχείριση για ποιο λόγο, διότι όχι μόνο ενισχύουμε την ευθύνη της ιδιοκτησίας των κρατών μελών, αλλά έχοντας δύο ταμεία και κοινή διαχείριση και αντί να έχουμε ε, ετήσια λήψη αποφάσεων, ε, να έχουμε ένα πολιετές πρόγραμμα, επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει μακροπρόθεσμη άποψη για το τι μπορεί να κάνει κάποιο κράτος με τα χρήματα τα οποία του διατίθενται. Από τις αρχές του 2013 θα έχουμε πολιτικό διάλογο με κάθε κράτος μέλος για να καθορίσουμε τους στόχους που θα καταρτιστούν για να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα προγράμματα που θέλουν να εφαρμόσουν και να συζητήσουμε τους στόχους τους οποίους επιζητούν και θα κατανέμονται οι πόροι αντιστοίχω. Ε, θα υπάρχει δηλαδή ένα πιο ευέλικτο σύστημα διαχείρισης των πόρων και όπως είπα στην απόφαση εδώ θα χρειάζεται ε, λιγότερο στρατηγικός προγραμματισμός. Οπότε αν και ε, εσείς και το Συμβούλιο υιοθετήσει την πρόταση το 13-14 θα είναι χρόνος εντόνων ε, συζητήσεων για να προγραμματιστεί το τι μέλη γενέστε και στον τομέα της ασφαλείας διότι για πρώτη φορά αντί να προτείνουμε ε, ε, να διαχειριζόμαστε μεμονωμένα θα τονίζουμε και στον τομέα της ασφαλείας την καταπολέμηση του ε, οργανωμένου εγκλήματος άλλων τομέων και ποιοι είναι οι πόροι που θα διατεθούν για αυτές τις δραστηριότητες. Θα υπάρχουν δηλαδή ε, πιο στρατηγική στόχη. Τι θα γίνει λοιπόν με το ποσοστό το οποίο θα παραμείνει στην κεντρική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα είναι να προωθήσουμε ε, τους διεθνείς στόχους. Υπάρχουν λίγες δράσεις οι οποίες είναι διεθνικές και υπάρχουν ε, ε, δεν υπάρχουν ε, κάθετες τομές αλλά οριζοντίως όταν πρόκειται για διεθνή φαινόμενα τα οποία καταπολεμούμε ή αλλού όπου στηρίζουμε ένα σύστημα επανεγκατάστασης και χρειάζονται πολύ περισσότεροι πόλοι για την επανεγκατάσταση ή όπου υπάρχει μία αποτελεσματική αποτελεσματική ε, χρήση των βέλτιστων πρακτικών, όλες αυτές οι ενέργειες οι οποίες θεωρούμε ενέργειες της ενώσεως θα παραμείνουν χρηματοδοτούμενος από το κέντρο με διαφορετικές τεχνικές και ε, μία από τις τεχνικές αυτές είναι σε συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις αλλά μία άλλη τεχνική είναι να χρησιμοποιούμε τα γραφεία μας όπως η Frontex και άλλα σαν οργανισμούς εφαρμοστικούς. Δηλαδή πέραν των χρημάτων τα οποία θα λαμβάνουν επιδοτήσεως για αυτές τις βασικές δραστηριότητες θα καθορίσουμε κατόπιν εντολής τους κατά περίπτωση πρωτοβουλίες όπου θα αναπτύσσονται και θα μπορούμε παραδείγματο χάρη εάν ε, χρειαστεί να συζητήσουμε με τις αρχές των τρίτων χωρών για να δούμε πόσο θα υπάρξει καλύτερη διαχείριση των συνόρων για να υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση αντί να χρηματοδοτούμε έναν σύμβουλο ο οποίος με τη συνήθη τεχνική ε, βοήθεια θα αναπτυχθεί θα αναθέσουμε στη Frontex να εκπαιδεύσει ε, ε, άτομα σε μία ευρωπαϊκή δράση που θα είναι συνεκτική θα έχει ολοκληρωμένο πλαίσιο και θα συμμετέχει σε ένα πλαίσιο που θα συνεργαστούμε με τη Europol, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα κράτη-μέλη κατά τρόπον ώστε η, η χρήση αυτή και η εφαρμογή να είναι κοινή και μπορούμε να αναφερθούμε και σε άλλες δραστηριότητες. Ένας ε, άλλος τρόπος ε, θα ήταν η πιο στοχευμένη χρήση της υπηρεσίας μας σε περιπτώσεις ad hoc για ιδιαίτερες περιπτώσεις. Υπάρχει επίσης το ζήτημα του καλύτερου εξοπλισμού για πιο γρήγορη επέμβαση σε περίπτωση εκτέκτης ανάγκης. Πιστεύω ότι όλοι παρατήρησαν κατά τα πρόσφατα επεισόδια ε, και των καταστάσεων κρίσης στα εξωτερικά μας σύνορα ότι οι δυνατότητε μα ε, κινητοποίησης χρημάτων γρήγορα για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη που βρίσκονται υποποίηση για να κινητοποιήσουμε όχι μόνο τις υπηρεσίες αλλά και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων είναι περιορισμένη. Γι' αυτό το λόγο θα θέλαμε να αυξήσουμε τα κονδυλία που μπορούν να αφιερωθούν σε ε, δράση έκτακτη ανάγκης ε, για πολύ πιο γρήγορη κινητοποίηση τη υποστήριξη. και επίση να έχουμε περισσότερα χρήματα αφιερωμένα σε δράσει σε τρίτε χώρε. Πολλές φορές εδώ έχουμε συζητήσει και επίση έχω ακούσει αρκετές ανησυχίες ε, ότι ο τομέας πολιτικής μας ε, που καλείται σε μεγάλο βαθμό να ε, παρέμβει εκτός των συνόρων μας για τη διαχείριση της μετανάστευσης ή της ασφάλειας δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένη διότι κάθε φορά χρειάζεται να κάνουμε ε, να χρησιμοποιήσουμε ποσά που χρησιμοποιούνται για άλλου στόχου, όπω για την ανάπτυξη. Πολύ συχνά, ορισμένε φορέ, συζητάμε για το πώ θα χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια για την ανάπτυξη, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για άλλου σκοπού, για την ανάπτυξη και όχι για εμά, για να συμπληρώσουμε αυτέ τι ελλείψει. Έχουμε λοιπόν συμπεριλάβει ένα κεφάλαιο στην πρότασή μα, στην νομική βάση και για τα ποσά που θα ε, αφιερώνονται σε δράσεις σε τρίτες χώρες ώστε να δώσουμε κίνητρα ε, για αυτό. Για παράδειγμα, διαπραγματευτήκαμε μια συμφωνία για μια εταιρική σχέση κινητικότητας. Πολύ συχνά οι δυνατότητες χρηματοδότησης τη ε, υπηρεσία απαιτείται κάποια υποστήριξη. Τώρα μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να παίρνουμε χρήματα για την ανάπτυξη, για παράδειγμα, από τα αναπτυξιακά ταμεία και αποφεύγοντας τον τεράστιο κατακαιρματισμό που τελικά δεν βοηθάει στην όλη κατάσταση. Ένα ποσό χρημάτων λοιπόν χρειάζεται αφιερωμένο στην ε, δράση σε τρίτες χώρες. Όλα αυτά σε πλήρη συντονισμό με τα χρήματα που δαπανώνται σε άλλους τομείς. Όλα αυτά έχουν συζητηθεί ευρέως επίσης ε, και με τους συναδέλφους μας ε, στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στην ε, Γενική Διευθύνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά ας πούμε της αρχιτεκτονικής, απλοποίηση, ιδιοταμία, πολίτης, ε, χρηματοδότηση, κατανομή κονδυλίων σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ιδέα της διαχείρισης των εξωτερικών ε, συνόρων με λιγότερο κατακαιρματισμένο τρόπο, με την παραχώρηση κονδυλίων σε κράτη-μέλη που πραγματοποιούν τη διαχείριση των ε, συνόρων εκ μέρου όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Και επίσης ε, κοινή διαχείριση και συγχρηματοδότηση μαζί με ένα κεντρικά διαχειριζόμενο ποσό για εκτακτές δόσει, ε, διακρατικά έργα και τρίτες χώρες. Και δηλαδή πιο στοχευμένη χρήση της υπηρεσίας μας. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική, έχει και οικονομικούς όρους, κάποια ευελιξία, από οικονομική άψη κάποια ευελιξία, ώστε αν τα ποσά για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης δεν χρησιμοποιηθούν πλήρως, να μπορούν να αναδιανεμηθούν στην κοινή διαχείριση. Προσπαθούμε λοιπόν να βελτιώσουμε την ευελιξία και να έχουμε τη μέγιστη φυσικά διαφάνεια ώστε να αξιοποιούνται πλήρως τα κονδυλία μας. Προβλέπουμε μία ενδιάμεση αναθεώρηση στη μέση της περίοδου ώστε να επαναξιολογήσουμε το τι έχει επιτευχθεί, να συμπληρώσουμε ενδεχομένω με κονδύλια, χρήματα που έχουν δαπανηθεί, οι περιπτώσεις ιδιαίτερη πίεση. Η κεντρική ιδέα είναι να είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι, πιο ευέλικτοι και πιο πολιτικοί στο διάλογο μας με τα κράτη-μέλη και λίγο λιγότερο να καθοδηγούμαστε από τον έλεγχο των τιμολογίων ως δραστηριότητα. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική. Τώρα, όσον αφορά τα κονδύλια τα ύψος των κονδυλίων που αποφάσισε να προτείνει η Κομισιόν στις ε, αρχές προπολογισμού, δηλαδή το Συμβουλίο και το Κοινοβούλιο, είναι 10,9 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2014-2020. Εδώ μιλάμε για καθαρή αύξηση περίπου 40% σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης περίοδου. Ωστόσο, ο υπολογισμός ε, δεν είναι απόλυτος. Ε, αποτελεί απλά αναφορά. Έχουμε πάρει το 2013 ως αναφορά, ως έτος δαπανών, διότι όπως γνωρίζετε ξεκινάμε λοιπόν με πολύ μικρά ποσά τα οποία αυξάνουμε για ποιο λόγο διότι την πρώτη φορά που η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη υλοποιούν δομημένη χρηματοδότηση σε αυτό το τομέα. Συνεπώς ε, αποφασίστηκαν οι δαπάνες σε πολύ χαμηλό επίπεδο και αυξάνονται όπου και το 2013 θεωρείται ότι έχουμε αποκτήσει τη σωστή ταχύτητα το ύψος ε, δαπανών έχει φτάσει σε ένα επίπεδο ρήμανσης. Έχουμε λοιπόν το φετινό έτος ως έτος 1, το αυξάνουμε κατά 1% και θα δούμε ότι σε σχέση με τα ποσά του 2013 υπάρχει μια συνέχεια. Εάν πάρουμε ωστόσο τα προηγούμενα ποσά και τα μελλοντικά, ε, βλέπουμε μια αύξηση 40%. Ωστόσο αυτό το 40% δεν έπεσε από τον ουρανό, δεν ήρθε από το πουθενά. Ε, δεν είναι κάποιος μαγικός υπολογισμός, είναι η πρόβλεψη της συνέχισης του επίπεδου του 2013 όπως προβλέπετε τώρα που θεωρείται ότι είναι το επίπεδο ορίμανσης τώρα η κατανομή αυτών των κονδυλίων μεταξύ των δύο ταμείων είναι ότι το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης προτείνουμε να λάβει 3,9 δις ευρώ και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας που καλύπτει επίσης και τα σύνορα 4,6 δις. Ε, έχουμε δηλαδή εδώ ποσοστό 35 προς 45%. Η αλλαγή σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι τα σύνορα αυτή τη στιγμή τα διαχειρίζεται το Ταμείο Ασφαλείας. Γι' αυτό λοιπόν παρατηρούμε αυτή την αλλαγή. Θα ήθελα απλά να επισημάνω, όπως είπα προηγουμένως, ότι στο εσωτερικό του κάθε Υπάρχουν κάποιες ειδικέ ανάγκες που επισημαίνονται. Θα ήθελα να επισημάνω ειδικότερα μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για το Κοινοβουλίο που είναι το resettlement, η επανεγκατάσταση. Επειδή το άσυλο λαμβάνεται... Έχουμε λάβει πολύ ε, υπόψη μας ε, Έχουμε αφιερώσει 560 εκατομμύρια στις για τις πρωτοβουλίες επανένταξης και ώστε εσείς να αποφασίσετε μαζί με το Κοινοβούλιο τις προτεραιότητες όσον αφορά την επανένταξη. Αυτό σας είπα όταν συζητούσαμε το ενδεχόμενο να βρούμε μια λύση τώρα. Αυτό προτείναμε και η Κομισιόν ε, το εγκρίνει. Ας ελπίσουμε ότι στο τέλος της διαπραγμάτευσης θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό ήθελα να επισημάνω πιο ειδικότερα επειδή το έχουμε συζητήσει πολύ εδώ. Προβλέπουμε ε, κίνητρα για το Ταμείο Ασφαλείας ώστε να, να υποστηριχθούν οι πέντε στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της σχετικής στρατηγικής. Τα έχουμε λοιπόν ως σημεία αναφοράς ώστε ε, φυσικά μπορεί κανείς να κάνει πολλά πράγματα αλλά εδώ έχουμε την εσωτερική ασφάλεια με πέντε προτεραιότητες οπότε τα λαμβάνουμε αυτά ως σημεία αναφοράς. Υπάρχει το ειδικό ζήτημα σε αυτή την περίπτωση της μελλοντική υπηρεσίας ε, εφαρμογών ε, πληροφορικής που σχετίζεται με κάποια ε, μελλοντικά έργανα όπως το πακέτο έξυπνων συνόρων που θα ανατεθούν σε αυτή την υπηρεσία. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πόσο εδώ που έχει δεσμευτεί ώστε να δείξουμε ότι όταν θα κάνουμε την πρόταση για αυτό το πακέτο έχουμε και τα αντίστοιχα χρήματα ένα δισεκατομμύριο εκατό εκατομμύρια για την υποστήριξή του σε περίπτωση που υπάρξει φυσικά θετική απόφαση διαφορετικά μπορούμε να ε, μεταβάσουμε αυτά τα χρήματα σε κάποιον άλλο στόχο όσον αφορά τις υπηρεσίες ε, και αυτό είναι το τελευταίο μου σημείο Όσον αφορά τις επιδοτήσεις προς ε, υπηρεσίες που στον τομέα της εσωτερικής ε, ασφάλειας, ε, ΣΥΠΟΛ, υπηρεσία ναρκωτικών, Frontex κτλ. Ένα συνολικό ποσό 1,6 δις. Αυτές είναι οι βασικές επιχορηγήσεις που σημειώνουν πρόοδο φυσικά για να ληφθούν υπόψη νέα καθήκοντα ειδικότερα τα νέα καθήκοντα της ε, Frontex που προκύπτουν από τον νέο κανονισμό για τη Europol για... και επίσης και για άλλες υπηρεσίες ε, για προγραμματισμό όπως ε, για παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εκπαίδευσης όλα αυτά τα κονδυλία ανήκουν σε αυτό το 1,6 δισεκατομμύρια Εάν υπάρξουν επιπλέον ανάγκες για ε, πράγματα που θα προκύψουν στο μέλλον, μπορούμε να ε, ζητήσουμε να προσθεθούν κάποια χρήματα για υλοποίηση έργων, όχι απλά για να αυξηθεί το ποσό αυτό. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο η, η γενική περιγραφή της πρότασής μας ε, και αυτό που αποφάσισε η Κομισιόν δεν είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε προβλέψει εμείς και όπως σας εξήγησα ήδη ε, ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις, ε, τώρα θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η τρέχουσα κατάσταση έχει όπως έχει. Πιστεύω ότι ήμασταν αρκετά μετριοπαθείς. Όταν το συζητήσαμε εσωτερικά πολύ εξεπλάγησαν που ήμασταν τόσο μετριοπαθείς. Διότι από πολιτική άποψη είμαστε υπερβολικά εκτεθειμένοι. Πιστεύω ωστόσο το σημαντικότερο κομμάτι το πακέτο δεν είναι μόνο τα χρήματα, αλλά η αλλαγή του τρόπου δαπανών διότι δεν έχει νόημα να ε, έχουμε πολλά κονδύλια, το ξοδεύουμε όλο μας το χρόνο για λογιστικά θέματα. Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος μας, αυτή είναι η μορφή της πρότασής μας, αυτά είναι τα κονδύλια και τώρα συζητήσουμε και οι διαπραγματεύσεις φυσικά θα διαρκέσουν πολύ και ας δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Μανσερβίζη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί πραγματικά ήταν πολύ διεξοδική αυτή η παρουσίαση των προτεραιοτήτων. Διαπίστωσα ότι ήδη μερικοί συνάδελφοι έσπευσαν να ζητήσουν το λόγο. Ο γύρο των ομιλητών ξεκινάει με τον κύριο Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Μασερβίζη για την ε, σαφέστατη και περιεκτικότητη παρουσίαση του ε, των σχεδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω τέσσερις ε, σύντομες παρατηρήσεις, αν επιτρέπετε. Καταρχήν, ε, μια γενική πολυθετική αντίδραση για τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα η δική μου ομάδα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θα ε, υπογραμμίσει κυρίως δύο σημεία. Καταρχήν, τα τα ταμεία που υπάγονται στην κεντρική διαχείριση και που θα έχουν την ελαστικότητα να αντιμετωπίσουν ε, ε, περιστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Αυτό είναι κέρια σημασία για μας, γιατί ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε και μια ανελαστικότητα, αλλά και έναν κατακαιρματισμό. Δύο παράγοντες που μας εμπόδισαν ε, να, αντιδράσουμε ταχαίως και να ανταποκριθούμε σε επίγουσες καταστάσεις. Αυτή λοιπόν η αποκατάσταση της ελαστικότητας μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος. Ένα άλλο σημείο αφορά το χρηματοδοτικό σκέλος, το, το χρηματοοικονομικό σκέλος της συνεργασίας μας ε, με τρίτες χώρες σε θέματα μετανάστευσης. Είπατε επανειλημμένως σε μιλή στην Επιτροπή μας, κύριε Μασερβίζη, ότι όταν έχετε διαπραγματεύσει με τρίτες χώρες για μεταναστευτικά ζητήματα, δεν έχουμε ε, αρκετά κίνητρα, δεν δίνουμε αρκετά ενάυσματα στις ε, χώρες ε, προκειμένου να δεχτούν τα αιτήματά μας για τη μετανάστευση. Δεν έχουμε αρκετή διαπραγματευτική ισχύ. Διαβεβαιώστε μας ότι αυτή η αδυναμία περιορίζεται στο παρελθόν και ως εκ τούτου τα κονδύλια που θα χρειαστούν για να ενισχύσουν τη συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης θα συμπεριληφθούν για να ενισχύσουν την ισχύ μας στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουμε ότι οι διαπραγματεύσει με τρίτε χώρες για τη μετανάστευση θα πρέπει να συνδέονται με τις ευρύτερε διαπραγματεύσεις και σε άλλα θέματα. Γιατί και εσείς επισημάνατε ότι είναι πολύ δύσκολο να δελάσουμε τρίτες χώρες να ενδιαφερθούν για τη μετανάστευση αν δεν υπάρχουν ε, στι διαπραγματεύσει και άλλα θέματα. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένας χρηματοοικονομικός και δημοσιονομικός σύνδεσμος, αλλά όχι μόνο ο οικονομικός. Σε ό,τι αφορά τη Frontex, δεν ε, είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα καλά. Τα 1,6 δισεκατομμύρια που προτείνεται ε, επιχορηγήσεις για τους οργανισμούς θα περιλαμβάνουν και τα κονδύλια ε, που θα προσθεθούν στον προπολογισμό της Frontex που θα έχει τώρα ευρύτερες αρμοδιότητες γιατί γνωρίζετε ότι μεταξύ άλλων η Frontex θα μπορεί να αγοράζει και τον τεχνικό της εξοπλισμό πια. Οπότε μας ενδιαφέρει η θέση σας ε, κατά πόσο θα αυξηθεί ο προπολογισμό και η Frontex έχει ήδη προγραμματίσει πώς θα αγοράζει το τεχνικό εξοπλισμό μέχρι το 2020 και τι θα γίνει με τη σχετική χρηματοδότηση. Τέλος, είπατε ότι το τμήμα της ασφάλειας, που θα είναι το 55% των συνολικών κονδύλιων, θα περιλάβει και χρηματοδότηση για μεθοριακή ασφάλεια, ασφάλεια των συνόρων, ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων. Και έτσι εξηγείται η διαφορά μεταξύ των δύο. Ήθελα μια διευκρίνηση για το σημείο αυτό. Γενικώ πάντως και περιμένοντας και τις ε, λεπτομέρειες της πρώτης στους επόμενους μήνες. Η αρχική μου αντίδραση είναι πολύ θετική για τα προγράμματα, τα χρηματοδοτικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Γιγιόμ, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, Γενικό Διευθυντή που μας παρουσίασε αυτή την αναδιάρθρωση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα χρηματοδοτικά προγράμματα στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων και είναι μια αναμενόμενη αναδιάρθρωση, ιδιαίτερα στο Ταμείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, για δύο κατηγορίες λόγων. Καταρχήν, ε, διαπιστώθηκαν κάποιες τις όπως επισημάνατε και εσείς ο ίδιος, ε, και αδυναμίες του ισχύου του συστήματος, κάτι που ε, κατέστησε κάτι που απαραίτητη αναδιάρθρωση και επίσης είπαμε ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις. Θα ήθελα να επισημάνω τέσσερις αδυναμίες που εντοπίσαμε. Καταρχήν, έλλειψη ελαστικότητας ορισμένων μηχανισμών κάτι που καθιστά δύσκολη την ε, προσαρμογή τους και η δυνατότητα ταχείας αντίδρασης σε περίπτωση κρίσης ή εκτάκτου ανάγκης κάτι που διαπιστώνουμε ότι υπάρχει συχνά. Επίσης είπατε ότι διαπιστώσατε και ανεπάρκεια αυτών των κονδύλιων, παρόλο που στις εσωτερικές υποθέσεις οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες όλο και ενισχύονται. Κάτι άλλο που διαπιστώνουμε είναι και μία απώλεια αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή των ετησίων προγραμμάτων, ενώ ο προγραμματισμός γίνεται πια σε πολυετή βάση. Και τέλος, κάτι που φαντάζομαι συνέτεινε στην ε, νέα πρόταση, είναι η περιπλοκότητα και το άχθος των διαφόρων διαδικασιών. Κάτι που έχει αντίκτυπο στη διαδικασία της πληρωμής, δημιουργεί καθυστερήσεις και δημιουργεί και προβλήματα στους ε, διαφόρους ε, φορείς των προγραμμάτων και τις μη οργανώσεις. Κάποιες αναδιαρθρώσεις μερικές φορές έχουν και πολιτικό αντίκτυπο. Θα πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε και να μεριμνήσουμε ώστε τα συμφέροντά μας σε θέματα ασφάλειας να μην υπερισχύσουν και να μην επισκιάσουν τις υπόλοιπες προτεραιότητες των ταμείων αυτών. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω έκκληση για να ε, ε, αποκατασταθεί μια ισορροπία ως προς την κατανομή. Και τέλος, ένας προβληματισμός. Αυτή η αναδιατύπωση το, της χρηματοδότησης δεν θα πρέπει να αποτελέσει έκφραση μιας συρρήκνωσης του προϋπολογισμού, ενός δημοσιονομικού περιορισμού. Και δύο τελευταία σχόλια. Τα μία αυτά θα πρέπει να εξασφαλίσουν και τα, κονδύλια, τα νέα κονδύλια να εξασφαλίσουν μια ταχεία αντίδραση στις κατεπίγουσες περιστάσεις. Γιατί γνωρίζουμε ότι καταστάσεις που αφορούν το άσυλο και τη μετανάστευση μπορεί να έχουν ραγδαίες εξελίξεις, όπως διαπιστώσαμε και τους τελευταίους μήνες. Και να επιμείνω στην ανάγκη αποτελεσματικότητας του πολιετούς προγραμματισμού, ώστε η διαχείριση να καταστεί όντως πιο αποτελεσματική. Σας ευχαριστώ κύριο Σταβάρης. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ μιλάμε για εργαλεία. Πιστεύω ότι αυτό που έχει σημασία για τη χρήση των εργαλείων είναι οι στόχοι για τους οποίους ε, τα χρησιμοποιούμε και τους οποίους επιδιώκουμε. Για να είμαι σαφής, αυτή δεν ήταν η κατεύθυνση που είχε το Κοινοβούλιο πριν από μερικά μόλις χρόνια στην ε, δική μου εκθέση για την επανένταξη, όχι μόνο εγώ συζητή, αλλά και το Κοινοβούλιο, ε, επιθυμούσαμε επιτάχυνση ε, διαχωρισμό του Ταμείου για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη σε διάφορα ταμεία ώστε να έχουμε ένα ταμείο ειδικό για την επανένταξη επειδή το πρόβλημα εδώ είναι ότι όταν έχουμε τεράστια χρηματικά ποσά δεν έχουμε αρκετή πνευματική ας πούμε, ιδιοκτησία και δημοκρατική ε, ε, ιδιοκτησία όσον αφορά τον τρόπο που αυτά θα δαπανηθούν. Το βήμα μας προτείνεται είναι ένα τεράστιο βήμα που θα αποτελέσει υπόδειγμα, παράδειγμα για το μέλλον. Δεν λέω ότι είναι λάθος επειδή το Κοινοβούλιο κινείται προς άλλη κατεύθυνση. Απλά αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι αυτά τα εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθεί η αξιοπιστία της διαδικασίας και η πολιτική ευφυΐα την οποία χρειαζόμαστε. Μου αρέσουν πολλά από αυτά που λέτε όσον αφορά τη μεγαλύτερη ευελιξία Ε, ορισμένα όμως άλλα πράγματα με ανησυχούν. Θα χρησιμοποιήσω το δικό μου τομέα ως παράδειγμα, αλλά είμαι βέβαιος ότι αυτό συμβαίνει σε όλους τους τομείς. Ε, πώς θα είμαστε βέβαιοι ότι οι στόχοι που επιθυμούμε να επιτύχουμε με το ειδικό ταμείο για την επανένταξη θα επιτευχθεί ούτως ή άλλως. Πώς ξέρουμε ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την επαναγκατάσταση. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα και έχουμε όλο και μεγαλύτερους ε, αριθμούς προσφύγων. Αυτός είναι ο στόχος. Και να δώσουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα στην επαναγκατάσταση. Μετά έχουμε την μονάδα επαναγκατάστασης. Εμείς ζητήσαμε να υπάρχει σε δική μας έκθεση πρωτοβουλίας Εδώ μιλάμε ήδη για... Είμαστε... Έχει ξεκινήσει σχεδόν το 2012 και δεν έχει προβλεφθεί τίποτα για μια μονάδα επανεγκατάστασης για το 2012, ίσως το 2013. Στο μεταξύ όμως η μονάδα επανεγκατάστασης θα αποτελούσε ένα κρίσιμο βήμα για να υπάρχει αυτή η διάκριση, αυτή η ευφύ, αυτός χρήση τρόπος χρήσης των κονδυλίων διότι στην επανεγκατάσταση αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο πολύ τα κονδύλια που αφαιρώνονται εκεί, αλλά οι ανθρώπινοι πόροι και το είδος και, κάποια... και το ποια αφοσι... πώς αφοσιωνόμαστε σε αυτό το τομέα. Από την άλλη πλευρά τα εργαλεία που προτείνεται είναι καλύτερα για την επίτευξη ευελιξίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Μία για την κοινή διαχείριση. Δεν ανησυχείτε για το τι θα συμβεί με την κοινή διαχείριση όταν τα κράτη-μέλη, ε, όταν ζητηθούν χρήματα στα κράτη-μέλη. και στην τρέχουσα κατάσταση μέτρων λιτότητας που και ότι οι στόχοι μπορεί να υποβαθμιστούν με αυτόν τον τρόπο. Οι στόχοι της Ένωσης που πιστεύω ότι είναι, είναι οι πιο ενδιαφέροντας, αλλά ποιος καθορίζει τι είναι στόχος της Ένωσης, ποια θα είναι η διαδικασία καθορισμού ενός τέτοιου στόχου. Θα προσπαθώ να είμαι σαφής. Εάν η είναι έτοιμη να καθορίσει στόχους της Ένωσης ε, ε, με δικές μας εκθέσεις πρωτοβουλίας ε, που ε, εμάς ως ε, φερέφωνα των Ευρωπαίων πολιτών δεν ξέρω κατά πόσο το Συμβούλιο θα συμφωνούσε με κάτι τέτοιο με ανησυχεί θέση του Κοινοβουλίου σε όλα αυτά πιστεύω ότι η ευελιξία είναι καλό πράγμα για την Κομισιόν αλλά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και πιο ευέλικτο τρόπο ελέγχου από το Κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να είναι κάτι που χρησιμοποιούμε μία φορά το χρόνο όταν συζητάμε για τον προπολογισμό. Ε, ολοκληρώνω σε ένα λεπτό. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε και πιο ευέλικτοι όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε αυτό αυτά τα νέα ευέλικτα και ευρύτερα εργαλεία που προτείνατε. Για να συνοψίσω, θυμάμαι τα λόγια του Αρτιέρο Σπινέλη όταν είπε ότι συνήθως οι άνθρωποι δίσταζαν αν θα προχωρήσουν με μια Ευρώπη διακυβέρνηση ή δημοσίων υπαλλήλων. Καλό είναι να έχετε τους δημοσίους υπαλλήλους, ως, ε, τους υπαλλήλους της ε, Ένωσης ε, ως, συναδέλφους σας, γιατί έχουν ευρύτερη άποψη. γνωρίζουμε τη διαφορά ένας καλός ε, υπάλληλος ο οποίος χρησιμοποιεί ε, σωστά την ευφυΐα του μπορεί να φέρει εκπληκτικά αποτελέσματα. Ο Αλτιερός Πινέλη είπε επίσης ότι δεν πρέπει να δίνουμε το βάρος μόνο στην Ευρώπη των ε, στελεχών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Μου αρέσει η ευελιξία Φανταζόμαι ότι τη χρειάζεστε, αλλά θεωρώ ότι χρειαζόμαστε ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ευχαριστώ κυρία Βίξτρομ. Συγγνώμη. Η κυρία Βίξτρομ, ε, εκπρόσωπος του της ομάδας Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σας συγχωρώ Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μασαρβίση, για την πολύ περιεκτική και ενδιαφέρουσα παρουσίαση και πολύ θετική και για μας. Θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι οι, τα θετικά όργανα ε, όταν προτείνουν κάτι έχουν υπόψη και την πολιτική βούληση και τις πολιτικές προθέσεις και συνέπειες. Αυτό είναι πολύ θετικό και μάλιστα σε περιόδους εκτάκτου ανάγκης ή σε απρόβλεπτες και φνηδιαστικές καταστάσεις είναι που υπάρχει πιο έντονο το αίτημα για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και για άμεση αντίδραση. Τότε στη, στην κρίση φαίνεται ο καλός καπετάνιος και φάνηκε ότι η εργαλειοθήκη μας ήταν πολύ κατακαιρματισμένη κατακαιρματισμένη. Τώρα φαίνεται ότι είναι πιο περιεκτική, πιο ελαστική και μπορεί αυτός ο μηχανισμός να κινητοποιηθεί πολύ πιο γρήγορα. Η εργαλειοθήκη όμως αυτή θα πρέπει να διορθώσει τις αδυναμίες ε, που παρατηρήθηκαν μέχρι τώρα για να ανταπεξέλθει στους στόχους της. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πιο ενεργό και πιο δραστήρια προσέγγιση και στο πρόγραμμά σας, στο σχέδιό σας που είναι πιο απλουστευμένο, πιο σύγχρονο και πιο ενημερωμένο και επίκαιρο. Ελπίζω να καταφέρουμε να αντιδράμε ταχύτερα αποτελεσματικότερα και αποδοτικότητα. Αν υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους και αν αυτό είναι και το ζητούμενο των νέων προτάσεών σα, τόσο το καλύτερο. Και ας μην ξεχνούμε ότι ακόμη και στα πιο θετικά σενάρια, το κοινό σύστημα ασύλου και μετανάστευσης θα λειτουργήσει με σωστό τρόπο. Εσείς πώς βλέπετε την προσαρμογή των δύο ταμείων ή την ε, λειτουργία των δύο ταμείων σε αυτό το νέο σενάριο με θέση σε ισχύ του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και Μετανάστευσης. Και μια τελευταία παρατήρηση. Ας μην ξεχνούμε και τη σημασία του δημοκρατικού ελέγχου, του κοινοβουλευτικού ελέγχου εν προκειμένου δηλαδή. Ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλο ενδιαφέρον σας ακούω πάντα κύριε Μανσερβίση και πάντα μαθαίνω πράγματα από τις παρουσιάσεις σας. Ωστόσο δεν άκουσα τίποτα σε σχέση με την αξιολόγηση των, ε, της χρηματοδότησης. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έλαβα μια απάντηση σε μια έγγραφη ερώτησή μου όσον αφορά την κατανομή κονδυλίων στο ΤΕΚΙ για τη συνεργασία του ΤΕΚΙ και απάντησα ότι 440 εκατομμύρια κατανέμονται στο ΤΕΚΙ έως το 2013. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η συνεργασία με την Τουρκία βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Εδώ μιλάμε για χρηματοδότηση της συνεργασίας με την Τουρκία. Πιστεύω ότι κανείς δεν είναι ικανοποιημένος με τη συνεργασία με την Τουρκία. Ωστόσο, για αυτό το στόχο ξοδέψαμε όλα αυτά τα χρήματα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ακούω ότι θα αυξήσουμε τη χρηματοδότηση για όλες αυτές τις διαστάσεις έως το 2020 αλλά τελικά το 2020 θα ξέρουμε κατά πόσο επιτέχθησαν τα σωστά αποτελέσματα με όλα αυτά τα κονδύλια που ξοδέψαμε. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βερζάτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Μανσαμπίνη διότι όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζεται περισσότερη συνοκτικότητα, περισσότερη και καλύτερη διαχείριση των πόρων και, να, και, και απάντηση στις επίγουσες καταστάσεις. Διαφωνούμε όμως ως προς την κατάρτιση προτεραιοτήτων μεταξύ των επιγουσών καταστάσεων διότι στα σύνορα της Ευρώπης έχουμε και συμφωνούμε όλοι. Αλλά ε, πρέπει να γίνει μία συζήτηση για τις αιτίες αυτών των διαφωνιών και όσον αφορά τη δικιά μου πολιτική ομάδα οι διαφωνίες αυτές οφείλονται στην έλλειψη αλληλεγγύης του συνόλου των κρατών μελών σε αυτό το θέμα. Δεν θα αναφερθώ εδώ ή στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίστηκε ε, τη, τους ε, μετανάστες από τη Λιβύη όταν ξεκίνησε ε, ο πόλεμος αλλά η ανάληψη από ένα κράτος μέλος αυτών των μεταναστών ε, ήταν μοναδική. Όταν λοιπόν ακούω ορισμένε κυβερνήσεις κρατών μελών οι οποίοι θέλουν να μειώσουν την τακτική μετανάστευση ενώ είναι μεταξύ αυτών που είναι οι λιγότερο αλληλέγγυοι ε, ε, όντας Γαλλίδα δεν θα επεκταθώ αλλά αντιλαμβάνεστε για ποιον μιλάω. Και εδώ θα αναφερθώ στο παράδειγμα της Frontex, διότι ε, πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ε, τον, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η ισορροπία ε, την οποία έχουμε επιτύχει δεν ε, ευνοεί τα δικαιώματα του ανθρώπου και θέλω να αναφερθώ τώρα στη σωτηρία στη θάλασσα είχαμε 2.000 νεκρούς ήδη τον Οκτώβριο εφέτος έναντι ολόκληρου έτους πέρυσι. Θέλω λοιπόν να κάνω μία ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του θέματος. Η απάντησή της δεν με ικανοποιεί γιατί παραπέμπει στα κράτη-μέλη. Το να σώσουμε ανθρώπινες ζωές πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας στα κατεπήγοντα. Όταν οι ανεπάρκειες των κρατών μελών είναι προφανείς, επί του θέματος τόσο όσον αφορά την ε, την υποδοχή ε, των, ε, μεταναστών που παραπέουν και πλέουν στη Μεσόγειο όσο και για την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τα ανθρώπινα δικαιώματα η οποία πρέπει να βελτιωθεί για να συζητάμε με τρίτες χώρες διότι αν δεν βελτιωθεί εικόνα αυτή δεν μας πιστεύουν οι και οι τρίτες χώρες. Ευχαριστώ. Κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον, τον κύριο Μαν Σερβίζη. Έφτασα κάπως καθυστερημένα αλλά έγκαιρα για να ακούσω τα υπόλοιπα σχόλιά σα, Άφησα όμως έμπιστους ε, συνεργάτες ε, που σημείωσαν ε, λεπτομεριακά την παρουσίασή σας. Πάντως έφτασα εγκαίρως για να ακούσω κάτι που με προβληματίζει και θα ήθελα κάποιες εξηγήσεις. Μιλήσατε για τα 1,6 δισεκατομμύρια της επιχορηγήσεις για τους οργανισμούς. Είπατε ότι λαμβάνονται υπόψη νέες αρμοδιότητες και εξουσίες της Frontex, το επισήμανε αυτό και ο Σάιμον, αλλά είπατε κάτι που με προβλημάτισε και με ανησύχησε. Είπατε ότι ε, με βάση τη νέα λισαβονοποιημένη νομική βάση και η Europol δικαιούται ένα ποσοστό από το 1,6 δισεκατομμύρια, αυτό το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων για τους οργανισμούς. Μια και δεν ξέρουμε ακόμη γιατί μιλάμε με ακρίβεια, γιατί ε, η Frontex και η νέα Frontex είναι πια πραγματικότητα, ενώ η Europol βρίσκεται ακόμη σε φάση ανεξάρτητης αξιολόγησης. Οπότε τι κριτήρια υπολογισμού χρησιμοποίησατε για αυτό το δημοσιονομικό κονδύλιο και, προς την, και για την Europol. Η νέα Ευρωπόλ θα αποτελέσει τον καρπό μιας συναπόφασης. Δεν θα είναι το αποτέλεσμα μιας μονομερούς απόφασης του Συμβουλίου, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα τι ποσοστό του 1,6 δισεκατομμύρια θα αφιερωθούν σε αυτή την φανταστική προς το παρόν Ευρωπόλ. Ο Κλοντ Μωράς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαντσιβίση για τις πολύ θετικές πτυχές της στρατηγικής ευελιξία, χρήση των ταμείων εκτεκτής ανάγκης λοιπά. Θέλω να τονίσω για μέρους της ομάδας μου το πραγματικό ζήτημα που θεωρώ που αφορά την όλη στρατηγική τι θέση ακριβώς θα έχει το Κοινοβούλιο. Όταν μιλάτε για τα δύο ταμεία, εάν πάρουμε για παράδειγμα το άσυλο και τη μετανάστευση, σαφώς ε, αυτός είναι τομέας υψηλά πολιτικός και υπάρχουν διαφορετικές προτεραιότητες ανάλογα με το κράτος μέλος. Μας ανησυχεί λοιπόν ότι με την κοινή διαχείριση θα έχουμε πολιτικές αποφάσεις που θα λαμβάνονται αλλά και πώς αυτές θα επηρεάσουν το στρατηγικό μας όραμα και σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας δεν μίλησαν πολλοί συνάδελφοι για τη στρατηγική θα πρέπει να δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ για το ποια θα είναι τα όρια μεταξύ οργανωμένου εγκληματό και τρομοκρατίας γιατί φυσικά το οργανωμένο όγκλημα, έγκλημα βρίσκεται υψηλότερα στην ε, ατζέντα μα. Ε, θα θέλαμε να μα δώσετε κάποια ιδέα για το τι θα γίνει στους επόμενους μήνες. Η κυρία Οσελίνο, παρακαλώ να είστε σύντομοι. Μία παρατήρηση. Μιλήσατε για κάτι σημαντικό. Υπάρχει μια πιο στρατηγική προσέγγιση και λιγότερο κατακαιρματισμένη. Από αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε για να έχουμε μια πιο σαφή άποψη του τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Γιατί ως μέθοδος φυσικά είναι σημαντική, αλλά θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά αυτή την προσέγγιση. Σήμερα το απόγευμα θα έχουμε την παρουσίαση από την Κομισιόν της Στρατηγικής για την Ευρώπη και έτσι θα δούμε πού βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά από την παρουσίαση του πρώτου εγγράφου και αυτό θα μπορέσει να μας κάνει να καταλάβουμε και τα, για τα πέντε σημεία που αναφέρει η Κομισιόν πώς μπορούμε να κατανέμουμε και να δράσουμε και πώς να κατανέμουμε τα ε, κονδύλια. Σε τι δίνουμε προτεραιότητα ανάμεσα σε αυτά τα πέντε σημεία επειδή αυτά δεν είναι ισότιμα Συμφωνώ με όσα υπογράμμισαν πολλοί συνάδελφοι. Χρειάζεται μέγιστος έλεγχος εκ μέρους του Κοινοβουλίου σε αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει οπωσδήποτε σε καταστάσεις τέτοιες να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Εδώ μιλάμε για πολυετή προγραμματισμό και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει ε, σε μεγάλο βαθμό τα κονδυλία αυτά και την ίδια στρατηγική. Ευχαριστούμε. Κύριε Μανσερβίση, επιστρέφουμε σε εσά. Έγιναν πολλές ερωτήσεις, μερικές μακροσκελείς. Αλλά κάντε ό,τι μπορείτε για να συνοψίσετε και έτσι να ε, ε, τηρήσουμε το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες σας, για τις ερωτήσεις σας που θα μας βοηθήσουν να διασαφηνίσουμε τι πρέπει να κάνουμε μέσα στους επόμενους μήνες πολλά θέματα εδώ αφορούν τη νομική βάση και θα δείτε ότι υπάρχουν άρθρα όπου αναφέρονται οι βασικοί στόχοι και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα διάλογο ο οποίος θα οδηγήσει σε ένα προγραμματισμό. Φυσικά αν είμαστε απόλυτοι ο διάλογος δεν θα έχει κανένα σκοπό. Δεν μπορούμε λοιπόν να δώσουμε όλες τις πληροφορίες σε αυτά τα έγγραφα. Αυτά τα έγγραφα αποτελούν μάλλον την αφιτηρία. Το σημαντικό είναι λοιπόν εδώ να αναγνωρίσουμε την αρχιτεκτονική, τα βασικά ποσά, τον τρόπο κατανομής, αλλά φυσικά σε αυτό το έγγραφο δεν θα βρείτε τι θα κατανομηθεί πού. Διότι εδώ απαντάμε σε ένα γενικό κανόνα, όπως για όλα τα δημοσιονομικά πακέτα, δηλαδή το να δώσουμε μία αφιτηρία. πολλά πράγματα θα χρησιμεύσουν για τη δεύτερη φάση. Αλλά στην πρώτη φάση πρέπει να αποδεχθούμε αυτή την πρόταση, διότι εδώ μιλάμε για κάτι που είναι πρόταση της Κομισιόν. Που για... Προτείνω λοιπόν να εργαστούμε σε αυτό, γιατί αν δεν έχουμε αυτό δεν ξέρουμε, δεν θα έχουμε κάτι να αντιμετωπίσουμε αργότερα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα την ερώτηση του κ. Μπουζουτήλ σε σχέση με τη σχέση μεταξύ της εξωτερικής χρηματοδότησης, θα έλεγα, και του ευρύτερου πλαισίου της διαπραγματεύσης διαφορών συμφωνιών. Αυτό που επιτυγχάνουμε εδώ είναι η αναγνώριση ενό αφούς πεδίου δράσης που θα ε, καθοδηγείται από την DG Home τουλάχιστον στους τομείς ε, πολιτικής αυτής της Γενικής Διεύθυνσης σε σχέση με το τι θα συμβεί. Αυτό που θα δείτε είναι ότι αυτά που θα υπάρχουν στον ε, εξωτερικό χώρο θα επικεντρώνονται σε δύο άξονες, ε, αναπτυξή πολιτική και πολιτική εταιρικών σχέσεων. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να δημιουργηθεί βάση συνοχής. Να συμπληρώσουμε δηλαδή κενά και όχι να αντικαταστήσουμε άλλους πόρους. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Σκοπός μας ήταν να προσθέσουμε κάτι το οποίο θα σχετίζεται άμεσα με την πολιτική διότι γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι και συχνά πόσο άδικο είναι να χρησιμοποιούμε ε, αναπτυξιακά κονδύλια για την πρόθεση άλλων στόχων. Φυσικά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο θα πρέπει επίσης να δούμε και την έννοια της αιρεσιμότητας εφόσον ισχύει. Στη δική μας πολιτική, στο δικό μας τομέα δεν μιλάμε μόνο για ανάπτυξη. Ε, η αιρεσιμότητα περιλαμβάνει περισσότερη κινητικότητα για περισσότερες διασφαλίσεις. Πώς μπορούμε να το επιτύχουμε λοιπόν το ζήτημα. Αυτό θα πρέπει να το εξετάζουμε για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Δεν μπορώ να σας δώσω δευτερεύοντα ποσά. Σας έδωσα ένα παράδειγμα για την ε, επανεγκατάσταση. Αυτά τα ποσά όμως δεν υπάρχουν, δεν υποδεικνύουμε τέτοια επιμέρους ποσά. Αλλά για τις εξωτερικές δαπάνες, σας είπα ότι για τις εξωτερικές δαπάνες αυτό που έχουμε εμεί στο νου μας ε, είναι μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι αρκετά χρήματα αυτά. Επαναλαμβάνω όμως ε, ότι δεν παρουσιάζουμε μια πρόταση διαρθρωμένη ε, βάσει συγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ξέρω κύριε Ράης ότι αυτή είναι διαρκώς η συζητήση μεταξύ ε, στελεχών του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Αυτό γίνεται σε όλους τους τομείς πολιτικής. Η απάντηση συνήθως είναι διαχείριση επικεντρωμένη περισσότερο στην πολιτική σημαίνει λιγότερη ε, ακαμψία, διότι αν προκαθορίσουμε τα πάντα ε, ίσως να εμφανιζόμαστε καλύτερα από πολιτική άποψη, αλλά αν μετά τα πράγματα δεν λειτουργήσουν σωστά, έχουν ξοδευτεί όλα αυτά τα χρήματα, δεν υπάρχει ευελιξία. Αυτό όμως είναι κάτι συνηθισμένο. Η συνηθιστές μα μας είναι να μην μπαίνουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Για να σας δώσω ωστόσο το παράδειγμα της ε, επανεγκατάστασης, αυτό που προτείνουμε εμείς, εάν κοιτάξετε το κείμενο, είναι συνδυασμό της υποστήριξης τη επανεγκατάσταση με δύο διαφορετικά μέσα. Το πρώτο είναι η βασική κατανομή ενός δεδομένου κράτου μέλου που θα υποστηρίξει τη διαδικασία και ένας φάκελος, ένα κονδύλιο κινήτρων που θα διανεμηθεί αργότερα βάσει συμφωνημένων προτεραιοτήτων για την επανεγκατάσταση σε ε, νοσιακό πλαίσιο και θα έχουμε συζητήσει με το Συμβούλιο και την Κομισιόν για να τα έχουμε καθορίσει και μετά θα τα συνδυάσουμε. Δεν θα πούμε στο κράτος μέλος τι θα κάνει, αλλά θα το θέσουμε όλο αυτό σε ένα πλαίσιο και βάσει των συζητήσεων που κάνουμε εδώ. Συνεπώς δεν χρειαζόμαστε όλες τις λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αυτή η προσέγγιση μας. Όσον αφορά τα κονδύλια για τους οργανισμούς που ανέφεραν πολλοί, Φυσικά κάναμε έναν υπολογισμό υπέρ της αύξησης για τους οργανισμούς. Το ε, κονδύλιό μας έχουμε λάβει υπόψη την ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη τι χρειάζεται η Frontex, τον νέο ρόλο της Europol και, της, και τον νέο ρόλο της EPOL. Ωστόσο, η Κομισιόν αποφάσισε να ομαδοποιήσει όλες τους οργανισμούς υπό την επικεφαλίδα 3 σε ένα ενιαίο κονδύλιο, το 1,6 δις. Έτσι έχουμε ένα ποσό το οποίο δεν έχει καθοριστεί για κάθε οργανισμό ξεχωριστά γιατί έτσι αποφάσισε η Κομισιόν. Αλλά τα ποσά που θα περιλαμβάνονται σε αυτό το 1,6 δισεκατομμύρια θα υπάρξει σημαντική αύξηση για τη Frontex διότι χρειάζεται να μπορέσουν να εκτελέσουν τις νέες τους, ε, τα νέα τους καθήκοντα. Για την Europol έχουμε κάποιες ενδείξεις. Ο ρόλος που παίζει ήδη η Europol ε, στη διαχείριση όσον αφορά τις τρίτες χώρες όταν θα έχουμε ίσως κάποιες PNR, TFTS, ε, όταν θα υπάρχει ένα σύστημα για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο Υπάρχει κάποια συμμετρία μεταξύ ε, πολιτικού και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού. Γι' αυτό προσπαθούμε ούτως ή άλλως να έχουμε κάποια αύξηση για τον καθένα από αυτούς τους ε, οργανισμούς. Πρωταγωνιστής των συζητήσεων στον προϋπολογισμό 2000 ε, η Frontex φυσικά θα απολαύει την αύξηση όπως είδατε και μετά η Σίπολ αλλά όλο αυτό θα εξερθούν από τις διαπραγματεύσεις. Προσπαθούμε να καλύψουμε τις νέες ανάγκες. Αλλά θα το δούμε το αποτέλεσμα όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Κυρία Γκυγιόμ, όσον αφορά το πολιετές δεν σας λέω ότι εδώ σας δίνω κάτι τέλειο απλά ξέρω από που ερχόμαστε και ε, είδα τι δεν έχουμε στη διάθεσή μας. Εάν θέλουμε να παρεύουμε γρήγορα σε όλα τα μέτωπα έχουμε μικρά περιθώρια τα οποία πρέπει να προσαρμόσουμε βάσει παράλογων διαδικασιών διότι κάθε φορά που αυξάνουμε κάτι είναι τέλειος παράλογο. Με ένα ποσό που διαχειριζόμαστε κεντρικά με τρόπο με τεχνικές γρήγορης κινητοποίησης ε, με τους διάφορους οργανισμούς. Αυτό τώρα ε, υπάρχει μέσα στο κείμενο. Θέλαμε να αποφύγουμε να καθορίσουμε ένα συγκεκριμένο ποσό διότι εάν δεν υπάρχουν περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αυτά τα κονδύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο. Το γεγονός ότι εμείς το αποφασίζουμε μέσω μιας κεντρικής δράσης θα πρέπει να ε, μας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε πιο γρήγορα αποφάσεις. Ε, δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρουμε. Ωστόσο, ο, δημοσιο... ο πολιετής προγραμματισμός που βασίζεται σε παρατηρήσεις των... Ο στόχος είναι να συνδεθεί αυτό περισσότερο με τους στόχους και λιγότερο με τις δράσεις και με τα έγγραφα. Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση στην ουσία. Η κατάσταση σήμερα είναι ότι τα κράτη-μέλη ε, επιχειρηματολογούν με το σκεπτικό ότι μου λείπουν τόσα και θα τα ζητήσω από την Ένωση. Μιλάμε εδώ δηλαδή για μία shopping list και όλα είναι δυνατά. Αφού κάθε, φορά, κάθε χρόνο αποφασίζουμε τι θα κάνουμε, εδώ μιλάμε για μία τεράστια χρηματοοικονομική διαχείριση. Μετατρέποντας τον προγραμματισμό σε πολυετή και έχοντας κοινή διαχείριση που συμμετέχει σε αυτό θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό να έχουμε, θα πρέπει να βασιστούμε σε διαφανή πολιτική συζήτηση επειδή όταν το κάθε κράτος μέλος θα μας λέει ότι θέλω τέτοιο αριθμό επανεγκαταστάσεων ε, ή θέλω τέτοιο αριθμό για το άσυλο και για τη μετανάστευση. Θέλω να υπάρχουν μαθήματα ή μαθήματα γλωσσών, όλο το πακέτο της ε, ένταξης. Θα τα βασίσουμε όλα αυτά σε στόχους και σε αποτελέσματα έτσι ώστε αντί να επιβλέπουμε μόνο τα δημοσιονομικά, να βλέπουμε και τι επιτυχάνεται με όλα αυτά. Και επιμένω στο ζήτημα της ασφάλειας, διότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όταν θα ρωτήσουμε κάθε κράτος μέλος ε, τι σκοπεύει να κάνει για παράδειγμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, τι δαπάνες ε, αφιερώνται σε αυτόν τον τομέα, εκεί θα μπορέσουμε να συγχρηματοδοτήσουμε. Ε, Εφαρμόζοντα όμω την κοινή διαχείριση σε όλα αυτά τα θέματα, ενθαρρύνουμε τα κρατημέλη να μα πούν ποια είναι τα σχέδιά του, για παράδειγμα, για την καταπολέμηση της, του οργανωμένου εγκλήματο, του σπόρου που θα αφιερώσουν σε αυτό. Το ίδιο και για την τρομοκρατία και έτσι θα συζητήσουμε με αυτού τη διάρθρωση του εγκλήματο στον χώρο κτλ. Το ζήτημα λοιπόν τη κοινή διαχείριση έχει ως στόχος ε, να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Εδώ δεν έχουμε διαφορετικούς κανόνες από αυτούς που εφαρμόζουμε σε άλλους τομείς ε, ε διαχείρισης. Θα υπάρξει κάποια αλληλεπίδραση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ακολουθεί τους κανόνες ε, της χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Θα κάνουμε ένα προγραμματισμό και μετά θα έχουμε μια πολιτική συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Οι κανόνες ε, της οικονομικής διαχείρισης είναι ότι η δέσμευση δική μας, όπως κάνουμε για το προγραμματισμό των αναπτυξιακών κονδυλίων, είναι να αναγνωρίσουμε τι πρέπει να γίνει και να έρθουμε εδώ να τα παρουσιάσουμε. Και να βεβαιωθούμε ότι ο διάλογος θα είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένος. Όσον αφορά τη συνεργασία με την Τουρκία, το ποσό που αναφέρατε, το οποίο διαχειρίζονται οι φίλοι μας από τις εξωτερικές υποθέσεις, γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοιο ποσό στον τρέχοντα προϋπολογισμό μας ε, για συνεργασία με την Τουρκία. Αυτά αφορούν την ΕΠΑ. Δεν ξέρω τι κάνουμε αυτό. Κάνουν πολλά πράγματα. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι καλύτερη συνεργασία με τους συναδέλφους μας που ασχολούνται με τη διεύρυνση, ώστε για παράδειγμα όταν εξετάζουμε το ζήτημα που αφορά το άρθρα 23-24 με τη διαχείριση των συνόρων θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα μακροπρόθεσμα βάσει της φιλοσοφίας των Ταμείων Προένταξης Αυτά τα ποσά είναι λοιπόν ακριβώς τα ίδια όσον αφορά την αξιολόγηση αξιολογήσαμε πολλά από τα κονδυλιά μας και άλλα κονδύλια αξιολογούνται όταν εγκριθεί αυτό το έγγραφο θα είναι πλήρες και θα έχει γίνει εκτίμηση αντικτύπου για την πρότασή μας. Θα το συζητήσουμε όλο αυτό για να σας δώσουμε περισσότερες ε, πληροφορίες. Τώρα, για το θέμα της Europol και της Frontex, κύριε Διασδεμέρα. Για τη Frontex υπάρχει αύξηση των κονδύλιων και προσπαθούμε να διαπιστώσουμε ε, ποιες είναι οι συνέπειες εφαρμογής ε, του αναθεωρημένου κανονισμού. Δεν θεωρούμε ότι Frontex αγοράσει σκάφη ή αεροπλάνα, αλλά ίσως ε, μισθώσει ή συνδιαχειριστεί ορισμένα πράγματα. Δεν πρόκειται να δοθούν υπέρογκα κονδύλια πάντως για το τεχνικό εξοπλισμό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προλάβουμε προγραμματίσουμε δράσει τη Europol. Πάντως η Europol κυρίως συνδέεται με επιχειρήσει και όχι με περιουσιακά στοιχεία τόσο. Μιλάμε περισσότερο για software, για λογισμικό, για κέντρα ε, κατά του εγκλήματο στον κυβερνοχώρο ή για βάση δεδομένων. Θέματα λογισμικού περισσότερο. Παρά. Πάντως δίκιο έχετε. Εμείς προτείνουμε ένα ποσό, ένα συγκεκριμένο κονδύλιο. Η για βαση δεδομενων θεματα λογισμικου περισσοτερο παρα δικιο εχετε συγκεντρώσει προτεινουμε ενα ποσο ενα συγκεκριμενο κονδυλιο η αποφαση τη ευρωπαικη Επιτροπή ήταν να συγκεντρώσει σε ένα μόνο ποσό μόνο ε, τις επιδοτήσεις και τώρα στις διαπραγματεύσεις θα δούμε τι μπορούμε να αφιερώσουμε σε αυτόν τον οργανισμό προκειμένου να ανταπεξέλθει στην αποστολή του. Πάντω, πολύ πιθανό. Αλλιώ υπάρχει κίνδυνο να μεταφερθούν κονδύλια από την υλοποίηση του ενό στόχου στον άλλον. Πάντω, όπω είδατε στο κείμενο, προσδιορίζουμε συγκεκριμένα κριτήρια για τις ε, για την εθνική κατανομή των κονδυλίων και φυσικά αυτά σχετίζονται με το στόχο και την πολιτική ε, πληθυσμό, έκταση κτλ. Αλλά λαμβάνουμε υπόψη και την έκταση των συνόρων, τα θέματα ασφάλειας, ε, την αέρια μεταφορά προκειμένου να δούμε πώς εντοπίσουμε τι επιχειρήσει και φυσικά μια τεχνική αντίστροφη με αυτή του ΑΕΠ προκειμένου να γίνει ο υπολογισμό. Όσο πιο φτωχή είναι μια χώρα, τόσο περισσότερα λαμβάνει ε, με βάση τον υπολογισμό μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, πιο στρατηγικές προτεραιότητες από τις πέντε. Η διαχείριση των συνόρων καλύπτεται πλήρω από ένα σημαντικό ποσό από την ασφάλεια και είναι ε, προφανές και βλέπετε τα κριτήρια στην κατανομή. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες προτεραιότητες ε, σχετίζονται με το διάλογο περιπολιτικής και με τους στόχους. Τώρα, η εργαλειοθήκη θα είναι κατανομή σε ένα κράτος μέλος, προσδιορισμός του τι θέλει να κάνει ε, το κράτος μέλος και διάλογος πολιτικής. Ε, πρακτική συνεργασία που προάγεται από, τον οργανισμό που λαμβάνει την επιδότηση και υπάρχουν και συγκεκριμένες δράσεις, δυνατότητα συγκεκριμένων συμβάσεων εφαρμογής μεταξύ οργανισμού και Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να αναλυθεί επιπλέον πρόσθετο έργο που σχετίζεται με συγκεκριμένη κατάσταση και το στοιχείο οι δράσεις που υπάρχονται σε κεντρική διαχείριση. Γιατί θέλουμε να δώσουμε και ενάυσματα για να γίνει πιο ορατή αυτή η προσπάθεια και φυσικά υπάρχουν και εξωτερικές σχέσεις. Αυτό είναι το γενικό αρχιτεκτόνημα, αυτή είναι η γενική δομή και θα δούμε αν θα καταφέρουμε να την εφαρμόσουμε, όχι μόνο για τις διαπραγματεύσεις για τα ποσά και την νομική βάση, αλλά και κατόπιν σε εφαρμοστικό στάδιο, αν όντως θα μπορέσουμε να την πραγματοποιήσουμε. Εδώ παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας, τις σκέψεις μας και μετά θα συνεργαστούμε για να τις υλοποιήσουμε. Αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι εγγυημένο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε για τις διεξοδικές σας ε, εξηγήσει ε, κύριε Μασερβίση. Ε, σας υπενθυμίζω ότι θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας στις 3 η ώρα με ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τη στρατηγική εσωτερική ασφάλειας. Ε, εκπρόσωπο και της Κόζη θα έχουμε. Η συγκεκριμένη κυρία Ρεταμπόρ Σαλίνο ε, παρακαλώ να επανέλθετε στην αίθουσα στις 3 για να συνεχίσουμε τις συνεδρία. Ευχαριστώ. Καλή σας όρεξη.